Συνάδελφοι, να ξεκινήσουμε τη συνεδρίασή μα. Σε ό,τι αφορά την ημερήσια διάταξη, θα ήθελα να σα προτείνω το εξή. Το πρώτο σημείο στην ημερήσια διάταξη, τη συζήτηση με τον Μπορί Τάρασουκ, τον οποίο γνωρίζουμε και από προηγούμενε συναντήσει και συζητήσει μα. Είναι ειδικό απασταλμένο τη Ουκρανική κυβέρνηση για θέματα τη Κρυμαία Νομίζω ότι είναι πραγματικά ο σωστός εταίρος μας για να συνομιλήσουμε. Ο συνάδελφος Γκάλερ συμφώνησε το σημείο το δικό του της ημερήσιας διάταξης ε, σε ό,τι αφορά την ε, συνάθρηση, την συνέλευση Ευρωπαϊκής Ένωσης Αφρικής. Να το συζητήσουμε αργότερα. Τον ευχαριστώ ιδιαίτερα. Δεν έχω ανακοινώσει να σας κάνω. Και περνάμε λοιπόν στο 4 της ημερήσιας διάταξης ανταλλαγή απόψεων με τον κύριο Μπόρις Τάρασεκ. Θα ήθελα να κάνω μία παρατήρηση αυτή εξ αρχή. Παρακάλεσα και καλωσόρισα τον κύριο Τάρασεκ για να μα παρουσιάσει την Ουκρανική τοποθέτηση σε ό,τι αφορά τι ε, εξέλιξει των τελευταίων του τελευταίου καιρού και θεωρώ ότι θα πρέπει να κάνει δηλώσεις και ανακοινώσεις επί του περιεχομένου. Καταρχάς λοιπόν με οποιαδήποτε ερμηνεία του διεθνούς δικαίου οι δράσεις της ε, Ρωσικής Ομοσπονδίας είναι αντίθετες προς το διεθνές δίκαιο. Κατά δεύτερον, συμμετείχα στη, λίγο στις ε, διασκέψεις των τριών υπουργών ε, εξωτερικών με τον τότε πρόεδρο Γιαννουκόβιτς και το πρώτο θέμα που αποφασίστηκε τότε ήταν εντός 48 ώρων να ε, τεθεί εκ νέου σε ισχύ το Συντάγμα του 2004. Δεν τήρησε όμως ε, τη δέσμευσή του ο πρόεδρος Γιαννικόβιτς και δεν υπέγραψε αυτή τη συμφωνία και δεν ε, ε εκπλήρωσε έτσι τις υποχρεώσεις του. Και απουσίασε λοιπόν και δεν τήρησε τη συμφωνία αυτή αυτό το, αυτή η απόφαση ήταν τμήμα της ε, Γενικότερης Συμφωνίας και γι' αυτό λοιπόν το Σύνταγμα αυτό σήμερα νομίμως έχει τεθεί σε ισχύ. Επίσης ε, στη Συμφωνία ορίζεται, ορίζονταν ότι εντός 10 ημερών θα εκλεχθεί από το Κοινοβούλιο νέα κυβέρνηση. Αυτό λοιπόν και έγινε βάσει της Συμφωνίας. Κατά τρίτον, το Κοινοβούλιο το οποίο έλαβε την απόφαση αυτή είναι το ερετό και νόμιμο κοινοβούλιο, το οποίο με συντριπτική πλειοψηφία ψήφισε για το Σύνταγμα αυτά και για, το, και την κυβέρνηση αυτή και για τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου. Άρα, όπως και να το ερμηνεύσει κανείς, Κατά τρίτον, λοιπόν, τους τελευταίους ε, μήνες παρευρέθηκα συχνά στην Ουκρανία και δεν ε, συναντήσαμε φασίστες στους δρόμους, αλλά άτομα που προσπίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα πολιτικά δικαιώματα. Και δεν είδα να υπάρχει διακριτική μεταχείριση του ρωσικού πληθυσμού. Και τα δύο λοιπόν στοιχεία είναι αυτά πράγματα και οι φασίστες και ε, η διακρατική μεταχείριση της ρωσικής ε, μειονότητας είναι στοιχεία τα οποία συστηματικά αναπτύσσει η ρωσική προπαγάνδα. Και γι' αυτό δεν υπάρχει οποιαδήποτε αντικειμενική βάση. Δεν μπορεί να υπάρξει λοιπόν επιχειρηματολογία. Σε ό,τι αφορά δηλαδή τους ε, ρωσόφωνους στην Ουκρανία και την ανάγκη υποστήριξής τους σε ό,τι αφορά δηλαδή Ουκρανούς πολίτες με ουκρανική υπηκότητα. Η νομοθεσία για τις ε, γλώσσες ποτέ δεν τέθηκε σε εφαρμογή, άρα ούτε αυτό το επιχείρημα στα Και άρα θεωρώ ότι τα αντικειμενικά ε, επιχειρήματα που μας προβλήθηκαν δεν στέκουν και ότι δεν πρόκειται παρά μόνο για μια πολιτική επίδειξη δύναμης για να συνεχιστεί η παράδοση της παλιάς αυτοκρατορίας. Αυτή είναι η δική μου ανάλυση της κατάστασης, το πώς θα το αντιμετωπίσουμε. Αυτό είναι το πιο δύσκολο τμήμα και νομίζω ότι θα πρέπει να το συζητήσουμε στη συνέχεια, αφόσον ακούσουμε και την άποψη του κυρίου Τάρασουκ για το πώς βλέπει την κατάσταση αυτός. Μπορείς, έχεις το λόγο. Thank you, Chairman. Thank you, Chairman. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Αγαπητά μέλη της Επιτροπής, είναι μεγάλη τιμή για μένα που μου δίνετε τη δυνατότητα να πάρω το λόγο εδώ. Θα ήλπιζα να σας μιλήσω και να σας ενημερώσω για την νίκη του λαού της Ουκρανίας πάνω στην δικτατορία που σοβούσε στη χώρα αυτή μετά από τρεις μήνες ειρηνικών διαπραγματεύσεων, ειρηνικών διαδηλώσεων, διαμαρτυριών μια μορφή αντίδρασης ε, στη στάση των Ουκρανικών αρχών να μην υπογράψουν τη Συμφωνία Σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για πρώτη φορά λοιπόν στην ιστορία της Ευρώπης ένας ολόκληρος λαός εξεγέρθη υπέρ των ευρωπαϊκών αρχών και των ευρωπαϊκών αξιών και οι αρχές ε, τελικά προσπάθησαν να καταστήλουν τις εκδηλώσεις αυτές με αποτέλεσμα 100 νεκρούς, 100 αθώους πολίτες οι οποίοι βία έχασαν τη ζωή τους, ήταν άμαχοι οι οποίοι δολοφονήθηκαν από ακροβολισμένους δολοφόνους και όλοι εμείς που για τρεις μήνες διαδηλώναμε στο Μαϊντάν Πιστέψαμε ότι έφτασε η στιγμή η Ουκρανία να πάρει την τύχη της στα χέρια της και να οδηγηθεί στην μεγάλη ευρωπαϊκή οικογένεια. Δυστυχώς όμως δεν συνέβη αυτό, γιατί μόλις, εξε, μόλις ήρθαν στην εξουσία οι νέες Ουκρανικές δημοκρατικές αρχές, η Ρωσία ξεκίνησε να εμποδίζει τον Ουκρανικό λαό να ζήσει το όνειρό του, να γίνει δηλαδή αναπόσπαστο τμήμα της ευρωπαϊκής κοινωνίας. Δεν θα ήθελα να σας μακρηγορήσω για την ιστορία ε, της Ουκρανίας τον τελευταίο καιρό. Θα ήθελα όμως να πω ότι είμαι εδώ μπροστά σας σαν ειδικό απεσταλμένος της Ουκρανικής κυβέρνησης για την ρύθμιση του προβλήματος της Κρυμαίας. Είναι η πρώτη μου μέρα που αναλαμβάνω αυτό το ρόλο. Είχα την δυνατότητα και στο παρελθόν να συναντηθώ με πολλούς από σας και ενθυμούμε με μεγάλη υπερηφάνεια ότι είχα υποδεχθεί και μία αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού ε, Κοινοβουλίου στο Μαϊντάν, στο λεγόμενο Euro Μαϊντάν και τους βοήθησαν να γίνουν κατανοητοί από τους διαδηλωτές. Όλες αυτές ήταν ιστορικές στιγμές και δεν πρέπει να ήταν ιστορικές μόνο για μας τους Ουκρανούς, αλλά και για σας, για τον κύριο Σαλαφράνκα, για τον φίλο Γιάτσεκ που ήταν στο Μαϊντάν και απευθύνθηκαν στους διαδηλωτές. Ένιωσα λοιπόν υπερήφανος γιατί είδαμε τι εγκαρδιότητα υποδέχθησαν οι διαδηλωτές τους εκπροσώπους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Εξέφρασαν την επιθυμία τους έτσι να γίνουν αναπόσπαστο τμήμα μιας δημοκρατικής μεγάλης Ευρώπης. Να σας υπενθυμίσω ότι αυτή στιγμή η νέα δημοκρατική κυβέρνηση ε, σχηματίστηκε την προηγούμενη Πέμπτη αμέσως δηλαδή μετά οι Ρώσοι άρχισαν τις δικές τους ενέργειες. Αυτό το οποίο στην παρούσα στιγμή συμβαίνει είναι το εξής. Με ρώτησε μάλιστα και ένας δημοσιογράφος ποια είναι η γνώμη μου για αυτό το οποίο κάνουν οι Ρώσοι. Έχουν εισβάλλει στην Κρυμαία ή όχι. Εγώ είπα ότι ήταν και ε, εισβολή και παρέμβαση στα εσωτερικά. Είναι διπλή η παρέμβαση η ρωσική δηλαδή. Κατά κάποιο τρόπο βέβαια ο τρόπος που έδρασαν οι Ρώσοι ήταν σε εισαγωγικά καινοτομικός. Στην ουσία παρενέβησαν με ένα συνδυασμό στρατιωτικών και πολιτικών μέσων ξεκίνησαν εισβάλλοντας στα κυβερνητικά κτίρια της αυτόνομης δημοκρατίας της Κρυμαίας. Δεν είχαν μαζί τους σημαίες, σήματα εθνικά. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο να φανήκαν ότι ήταν Ρώσοι αυτοί οι οποίοι εισέβαλαν στα κυβερνητικά κτίρια. 6.000 ειδικέ δυνάμεις εισέβαλαν στην Κρυμαία ε, η Κρυμαία είναι ένα απόσπαστο θυμίζω τμήμα του Ουκρανικού εδάφους. Η νέα κυβέρνηση έδωσε διαταγή στους στρατιωτικούς μας στην ε, Κρυμαία να μην ανταποδώσουν ε, πειρά, να μην δώσουν άλοθη στους Ρώσους, να μην δημιουργηθεί προβοκάτσια. Αντίθετα είδαμε τους Ρώσους οι οποίοι με κοινικό τρόπο μέσω των ειδικών δυνάμεων της μονάδας GRU, δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε τι είναι αυτή η μονάδα. Είναι μια μονάδα που εξαρτάται άμεσα από τις υπηρεσίες αντικατασκοπίας της τέος Σοβιετικής Ένωσης και τώρα της Ρωσίας είναι ειδικέ όπως είπαμε δυνάμεις για υπόγειες παρεμβάσεις, ανορθόδοξες μορφές πολέμου κτλ. Και χωρίς να φέρουν κανένα σήμα, χωρίς να φαίνεται ότι ανήκουν σε στρατιωτικές δυνάμεις ή ασδήποτε χώρας. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν 6.000 από αυτούς κατέλαβαν όλες τις κρατικές υπηρεσίες της Κρυμαίας και τερματίζουν όπου να είναι την επιχείρησή τους ελέγχοντας και διάφορες επιμέρους στρατιωτικές εγκαταστάσεις της Κρυμαίας. Θα ήθελα εδώ να υπογραμμίσω ότι ο Ουκρανικός στρατός στην Κρυμαία δεν χρησιμοποίησε το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει όπλα μετά από οδηγίες ή ουδήποτε. Η κυβέρνηση τους είχε πει μην χρησιμοποιήσετε τα όπλα σας. Φυσικά αυτές οι στρατιωτικές ενέργειες συνοδεύθηκαν και από πάρα πολλές προκλητικές πολιτικές παρεμβάσεις. Οι Ρώσοι αμέσως μετά την απόφαση της νόμιμης θυμίζω Βουλής του Κιέβου αμέσως είπε ότι δεν αναγνωρίζει τις νέες Ουκρανικές αρχές. Είπε ότι ναι μεν ήταν νόμιμα εκλεγμένο το Ουκρανικό Κοινοβούλιο και η κυβέρνηση η οποία είχε ψηφιστεί στο παρελθόν από εδώ και πέρα δεν είναι νόμιμη εκπρόσωπη. Προετοίμασαν λοιπόν την κοινή γνώμη, ε, προετοίμασαν ουσιαστικά την παραπλάνηση της κοινή γνώμης ε, μέσα από, τα, από την ενημέρωση, από τα μέσα ενημέρωσης, <coughs> λέγοντας ότι δεν αναγνωρίζουν τις Ουκρανικές αρχές, λέγοντας ότι οι Ουκρανικές αρχές είναι εχθρικές απέναντι στους ρωσόφωνους της Κρυμαίας και στην υπόλοιπη νότιο-ανατολική ε, Ουκρανία, κάτι το οποίο είναι απολύτως ψευδές. Διότι αν πάει κανείς και δει το τι συμβαίνει στο Κίεβο και στις άλλες μεγάλες πόλεις της Ουκρανίας, εύκολα θα καταλάβει ότι πολλοί κόσμος, οι περισσότεροι σε κάποιες περιοχές ομιλούν τη ρωσική. Κανένας λοιπόν δεν μπορεί να πει ε, αληθώς ότι οι Ρώσοι δεν ομιλούν τη δική τους γλώσσα. Και τώρα ακούμε και στη ε, ρωσικά μέσα ενημέρωσης ε, πολλούς ρωσόφωνους να διαμαρτύρονται για τη ρωσική παρέμβαση. Ρωσόφωνοι Ουκρανοί οι οποίοι διαμαρτύρονται για την στρατιωτική επέμβαση και την κατοχή ε, του τμήματος αυτού του Ουκρανικού εδάφους. Λοιπόν, αυτή ήταν η προσπάθεια των Ρώσων, πολιτικο-στρατιωτική στην ουσία χρησιμοποίησαν τις ε, δυνατότητες που είχαν στην Κρυμαία, οργάνωσαν εξεγεύσεις πολιτικού τύπου και παρενέβησαν. Ε, έδειξαν και διάφορα σκέτ στην τηλεόραση που δήθεν ήθελαν να αποδείξουν τα λεγόμενά τους, αλλά δεν υπήρξε ούτε ένας νεκρός και μόνο κάποιοι καμοφλαρωσμένοι Ρώσοι στρατιώτες περιπολούσαν εξοπλισμένοι σαν αστακοί στις πόλεις της Κρυμαίας όπως τη Συμφερόπολη και τη Σεβαστούπολη. Λοιπόν έτσι είναι δυστυχώς η κατάσταση. Θα πω εδώ ότι οι Ουκρανικές αρχές δεν έδωσαν κανένα λόγο, δεν προκάλεσαν κανέναν, δεν πυροβόλησαν κανέναν, δεν χρησιμοποίησαν καθόλου όπλα. Εμείς ελέγχουμε τις αντιδράσεις μας Ταυτόχρονα όμως η Ουκρανική Βουλή η οποία εργάζεται ε, συνεχώς, συνεδριάζει συνεχώς, κάνει ό,τι μπορεί έτσι ώστε να αποκατασταθεί η ειρήνη και να αποκατασταθεί η τάξη στην Κρημαϊκή Χερσόνησο. Εμείς μεταφέρουμε την έκκληση της Ουκρανικής Βουλής και στις εγκύτριες δυνάμεις, ιδιαίτερα μετά από την συμμετοχή της Ουκρανίας στην Διεθνή Σύμβαση για τη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων και μετά από την απόφαση της Ουκρανίας να καταστρέψει το σύνολο του πυρηνικού εξοπλισμού της. 176 διπυρωτικοί βαλιστικοί πύραυλοι και 2.000 πυρηνικές κεφαλές. Εγώ προσωπικά ήμουν πάρα πολύ κοντά στα πλαίσια της ε, υπογραφής αυτού του μνημονίου εγγυήσεων για την εθνική ασφάλεια. Θα ήθελα να πω ότι σε καμία περίπτωση δεν χρησιμοποιήθηκε το έγγραφο αυτό για την προάσπιση των Ουκρανικών συμφερόντων ούτε το 2003 όταν υπήρξε το πρόβλημα στο στενό Κέρτς, ούτε και τον προηγούμενο Αύγουστο όταν οι Ρώσοι στην ουσία επέβαλαν ε, εμπορικές κυρώσεις και έναν ιδιότυπο εμπορικό ε, αποκλεισμό. Το μνημόνιο της Βουδαχέστης προβλέπει δύο περιπτώσεις όπου θα πρέπει να τεθούν σε εφαρμογή οι εγγύησεις Μία περίπτωση. Όταν υπάρχει χρήση βίας ή απειλή χρήση βίας κατά της ε, Ουκρανίας, κατά της εδαφικής της ακεραιότητας και κυριαρχίας και δεύτερη περίπτωση εάν υπάρχει χρήση οικονομικών μέσων για να υπονομευτεί η οικονομία της Ουκρανίας. Και τα δύο αυτά λοιπόν στοιχεία θα έπρεπε να αντιμετωπιστούν στις διαβουλεύσεις. Για πρώτη φορά τώρα το μνημόνιο της Βουδαπέστης θα αρχίσει να λειτουργεί. Σήμερα στο Κιέβο έχουμε τον εκπρόσωπο του Ηνωμένου Βασιλείου, τον Υπουργό Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου, που είναι μία από τις εγκύτριες χώρες για το μνημόνιο της Βουδαπέστης. Αύριο θα είναι ο Υπουργός Εξωτερικών Κέρι των Ηνωμένων Πολιτειών, που και οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι εγγυητής αυτής της συμφωνίας της Βουδαπέστης. Σε ό,τι αφορά τους Ρώσους, οι Ρώσοι εξακολουθούν να αρνούνται να συμμετάσχουν στη συζήτηση ως μία από τις εγκύτριες χώρες για το μνημόνιο της Βουδαπέστης. Δεν θέλουν να έχουν ούτε διμερείς διαπραγματεύσεις και διαβουλεύσεις, ούτε υπό την ιδιότητά τους ως εγγυητές του μνημονίου της ε, Βουδαπέστης. Αυτό σημαίνει ότι δεν σέβονται ούτε τις ε, διεθνείς, τα διεθνείς συμφωνίες και τους κανόνες του διεθνούς δικαίου, ούτε τη χάρτα των Ηνωμένων Εθνών, ούτε την σημαντική διμερή συμφωνία που έχουμε κάνει μαζί τους, η οποία προβλέπει την ε, αμοιβαία υποστήριξη της εδαφικής ακεραιότητας της Ουκρανίας και της Ρωσίας και επίσης θέλω να σας υπενθυμίσω ότι εγώ ήμουν αυτός ο οποίος ξεκίνησε την ε, έγκριση του ενιαίου αυτού εγγράφου στις 20 Ιουλίου 1993, το εγγράφο αυτό που προετοιμάστηκε από το Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, που ενώπιον σε προκλητικής απόφασης του Ρωσικού Κοινοβουλίου κατά της εδαφικής ακυρεότητας της Ουκρανίας, ε, είπε το έγγραφο αυτό και ήταν απόφαση του ΟΗΕ ότι αυτή η δήλωση της Ρωσίας ήταν απόλυτα άκυρη και χωρίς περιεχόμενο και στρεφόταν εναντίον της χάρτας των Ηνωμένων Εθνών. Αυτό το έγγραφο παραμένει στη μέση διάταξη του Συμβουλίου Ασφαλείας και επομένως θα πρέπει να ληφθεί υπόψη αυτή η απόφαση. Είχαμε τις ε, συναντήσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας τις τελευταίες μέρες στη Νέα Υόρκη σχετικά και με αυτό το θέμα. Τι προσδοκούμε τώρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Φυσικά περιμένουμε την αλληλεγγύη σας όπως το έχετε τονίσει και κατά τη διάρκεια των τριών μηνών ειρηνικών διαδηλώσεων όταν οι διαδηλωτέ τονίζανε ότι θέλουν να είναι κομμάτι τη οικογένεια των Ευρωπαϊκών Εθνών. Τι χρειαζόμαστε όμω τώρα, χρειαζόμαστε κάτι περισσότερο από μία έκφραση αλληλεγγύης και δηλώσεων ε, υποστήριξης. Η εδαφική εκαιρεότητα και η κυριαρχικότητα της Ουκρανίας είναι σε κίνδυνο. Η Ρωσία ακολουθεί μια επιθετική πολιτική και έχει κάνει εισβολή σε ένα τμήμα του εδάφους μας. Έχουν παραβιάσει τις υποχρεώσεις τους ως συμβαλόμενοι για τη συμφωνία για την προσωρινή, ε, προσωρινό ελιμενισμό του ρωσικού στόλου στο έδαφος της Ουκρανίας. Αν πάρετε λοιπόν όλα αυτά τα έγγραφα στα οποία ε, είναι συμβαλόμενο μέρος η Ρωσία, όλα αυτά τα έγγραφα έχουν παραβιαστεί σε σχέση με τι υποχρεώσει που δεσμεύουν τη Ρωσία. Ελπίζουμε λοιπόν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πάρει ταχύτερα να το μια πολιτική απόφαση ώστε να υπογραφεί η Συμφωνία σύνδεση με την Ουκρανία, κάτι το οποίο οι προηγούμενε αρχέ τη Ουκρανία δεν υπέγραψαν, δεν δέχτηκαν να υπογράψουν και εξαιτία του οποίου έγιναν οι στην πλατεία Μαϊδάν. Είναι λοιπόν η προσδοκία μα ότι θα λάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή την απόφαση το ταχύτερο δυνατό. Η κυβέρνηση τη Ουκρανία είναι έτοιμη να προχωρήσει στην υπογραφή αυτή τη συμφωνία. Και παρενθετικά αυτή η συμφωνία ήταν πράγματι έτοιμη να υπογραφεί στις 29 Νοεμβρίου στο Βίλνιους. Ελπίζουμε λοιπόν ότι θα έχουμε την υποστήριξή σας για να γίνει αυτό πραγματικότητα. Και επίσης χαιρόμαστε για τις δηλώσεις οι οποίες προήλθαν από τους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά δεν υπαρκούν. Η τωρινή κατάσταση απαιτεί μία όχι παραδοσιακής μορφής απόφαση. Χρειάζεται μία πιο αποφασιστική στάση από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πιστεύω ότι θα ήταν σωστό η Ευρωπαϊκή Ένωση να αποφασίσει να δημιουργήσει μία ε, αποστολή παρακολούθησης της εξακρίβωσης σε σχέση με το τρόπο που μπορεί να παρακολουθηθεί η κατάσταση με τους συνοριοφύλακες της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι θα μπορούν να παίξουν κάποιο ρόλο αντίστοιχο με αυτό που διαδραματίζουν στην ε, Μολδαβία μεταξύ Μολδαβίας και Υπερνηστερίας. Πιστεύουμε λοιπόν ότι αυτός ο μηχανισμός από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα μπορέσει να αποδειχθεί ιδιαίτερα χρήσιμος. Αγαπητοί φίλοι, ως ε, συμπέρασμα θα ήθελα να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου σε όλους σας και ιδίω σε εσά που ήρθατε στην Ουκρανία κατά τη διάρκεια της πολιτικής κρίσης που αντιμετώπισε η χώρα μας. Όλοι εσείς που λάβατε το λόγο ενώπιον των διαδηλατών στο Μαϊδάν, νομίζω το καταλάβατε και ήδη, ακούσατε τον νιώσατε τον ενθουσιασμό του λαού μας που υποστήριξε εσά ως εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σας παρακαλώ να συνεχίσετε την υποστήριξη αυτή με συγκεκριμένα μέσα και τρόπους. Ευχαριστώ. Αγαπητοί συνάδελφοι, 14 ε, βουλευτές έχουν ζητήσει το λόγο. Σας παρακαλώ να συμφωνήσετε να πάρουν οι εκπρόσωποι των ομάδων δύο λεπτά και οι υπόλοιποι ομιλητέ ένα λεπτό. Και σας παρακαλώ όλοι να παραμείνετε σε, στο χρόνο αυτό ομιλίας ώστε στις 4 να μπορούμε να τελειώσουμε αυτή τη συζήτηση γιατί ο κύριος Τάριας πρέπει να μιλήσει και στα μέσα ενημέρωσης. Κύριε Σαλαφράγκα, έχετε το λόγο πρώτα. Όχι. Κύριε Τάριτ, μια διαδικαστική παρέμβαση. Είσαστε σίγουρος κύριε Πρόεδρε ότι όλες οι πολιτικές ομάδες είναι ενήμερες για αυτή τη συνάντηση γιατί κάποιες πολιτικές ομάδες δεν εκπροσωπούνται εδώ. Το γνωρίζουν. Κάποιες είναι πιο πληροφορημένες για την ένταση της πληροφορήσεως, λέει ο κύριος Μπρόκ. Κύριε Σαλαφράγκα. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Ταρασιούκ, καλώς ήλθατε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ζητήσατε αλληλεγγύη από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα ήθελα εξ ονόμα της ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος να εκφράσω την πλήρη μας αλληλεγγύη με σας και να καταδικάσω απερίφραστα τη ρωσική εισβολή στη χώρα σας. Θεωρούμε ότι μια πράξη που παραβιάζει το διεθνές δίκαιο και τη χάρτα των Ηνωμένων Εθνών και θέτει σε κίνδυνο την ε, ασφάλεια και την ειρήνη σε διεθνές επίπεδο. Είναι παράδοξο ότι μία από τις χώρες που είναι εγκύτριες για το μνημόνιο της ε, Βουδαπέστης που προστατεύει την εδαφική σας ακαιρεότητα είναι μια χώρα η οποία μετά από όσα έχουν γίνει στη Συρία ε, και όπου ζήτησε το Συμβούλιο Ασφαλείας να πάρει πρώτα απόφαση, τώρα παραβιάζει αντίστοιχε αποφάσεις. Επίκειται η συζήτηση και η απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας για την Ουκρανία και θα ήθελα να ξέρω κατά πόσο η κυβέρνησή σας, μετά από αυτά που είπατε για τη Συμφωνία Σύνδεσης, αν περιμένετε από την Ευρωπαϊκή Ένωση να προβούμε σε οικονομικές και πολιτικές κυρώσεις κατά της Ρωσίας και αν το Κοινοβούλιο σας ζητά το, συζητά το ενδεχόμενο να ζητήσετε να ενταχθείτε στο ΝΑΤΟ. Εκτιμούμε πολύ θετικά τις ε, ε, εντολές που έδωσε η κυβέρνησή σας να μην χρησιμοποιήσετε βία και να, ε, και να υπάρξει αυτοσυγκράτηση για να αποφευθεί μια σύγκρουση. Νομίζω ότι κανείς δεν θέλει τον πόλεμο, αλλά μέσα στο πλαίσιο στο οποίο βρισκόμαστε, κύριε Πρόεδρε, νομίζω ότι κανείς δεν μπορεί να ματαιώνει ε, για πάντα τις ε, προσδοκίες ενός λαού. Πάνω από 100 άτομα έχουν πληρώσει με τη ζωή τους αυτή την προσπάθεια να υπάρξει δημοκρατία στην ε, Ουκρανία. Πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να αρθεί στο ύψος των περιστάσεων. Δεν μπορούμε να παραδεχτούμε και να αποδεχτούμε μια τέτοια πράξη βαρβαρότητας που είναι η εισβολή σε ένα κυριαρχό κράτος. Um, thank you very much. Η κυρία Μποσκούρτ, σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την εισαγωγή σας, κύριε Ταρασίκ. Βλέπουμε μια κατάσταση η οποία διαρκώς κλιμακώνεται. Έχω κάποιες ερωτήσεις προς εσάς, γιατί είστε και ειδικός ε, απεσταλμένος για θέματα Κρυμαίας. Όπως ξέρουμε όλοι, την ε, Πέμπτη 50 ένοπλοι εισέβαλαν στο Κοινοβούλιο της Κρυμαίας. Και σύμφωνα με τις πληροφορίες που λάβαμε, μόνο τα μέλη της ε, ρωσικής ε, αντιπροσωπείας ε, μπορούσαν να εισέλθουν στο κοινοβούλιο. Οι υπόλοιποι έμειναν απ' έξω. Και αυτό που λέγεται είναι ότι η αστυνομία δεν ελέγχει την κατάσταση. Όταν λοιπόν ειδικό απεσταλμένο, ποιοι είναι οι συνομιλητέ σα, γιατί ελήφθη μια απόφαση βάσει δημοψηφίσματο την Πέμπτη και κατά δεύτερον ο Πρωθυπουργό καθαρέθηκε και αντικαταστάθηκε. Ποιοι είναι λοιπόν οι συνομιλητέ σα στην Κρυμαία. Κατά δεύτερον, για τα δικαιώματα των μειονοτήτων. Προφανώ υπάρχει μια μειονότητα 25%. Ουκρανοί και 15% Τατάρι των, ε, της Κρυμαίας οι οποίοι και διαδηλώνουν υπέρ της ενότητας και της ε, ακυρεότητα της Ουκρανίας και θα πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να τους βοηθήσουμε και να προασπίσουν με τα δικαιώματά τους. Τελευταίο σημείο. Ζητήσατε να υπογραφεί μία συμφωνία εταιρική σχέσης. Τι θα γίνει όμως μετά την υπογραφή αυτή, γιατί και αυτό ενδεχομένως να κλιμακώσει την κατάσταση. Ποια είναι η τοποθέτησή σας. Ο πρόεδρος Μπροκ, ήθελα να σας ενημερώσω ότι ο, ο πρωθυπουργός Άζαροφ ε, καθαρέθηκε και αποχώρησε υπό το Γιαννουκόβιτς και μετά ε, εκλέχτηκε νέος ε, πρωθυπουργός. Έτσι έγιναν τα πράγματα αντικειμενικά. Αυτά ήταν τα περιστατικά και τα γεγονότα. Ο κύριος Νταφ. Σας ευχαριστώ πρόεδρε. Εξ ονόματος των φιλελευθέρων θα ήθελα να εκφράσω την αλληλεγγύη μου Ο κύριος Πούτιν δρά σαν Ρώσος τύρανος. Φαίνεται ότι αντιδρά. Θα πρέπει να κατανοήσει ότι στο σύγχρονο κόσμο εξαρτάται από το παγκόσμιο οικονομικό σύστημα και από τις παγκόσμιες αγορές. Είναι πολύ πιο αδύναμος, πιστεύω, από ό,τι ενδεχομένως θεωρεί ή από ό,τι ενδεχομένως νιώθει. Υπάρχει λοιπόν μεγάλη περίπτωση επιβολής ε, σκληρών κυρώσεων, σε συνδυασμό και με την ανάγκη εντατικής άσκησης διπλωματίας. Θεωρώ ότι το ΝΑΤΟ έχει ένα πολύ μεγάλο πολιτικό ρόλο να διαδραματίσει εδώ, επιβεβαιώνοντας τους στόχους του και τη συνοχή του. Είναι κρίσιμη σημασία επίσης η Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι πολύ πιο σαφής και πολύ πιο ενωμένη. από ό,τι ήταν στο παρελθόν σε παρόμοιες κρίσεις. κατανοώ και δέχομαι την ανάγκη για έντονη παρακολούθηση των συνόρων και συλλογή μυστικών πληροφοριών. Ευχαριστώ. Η κυρία Μπόσκορτ. Τη ζητώ συγγνώμη, κατάλαβα λάθος αυτό που είπατε. Ε, νόμιζα ότι αφορούσε τον Πρωθυπουργό της Κρυμαίας. Αυτό που είπε ο κύριος Σόλτς έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Ταρασφιούκ, σας ευχαριστώ για την έλευσή σας εδώ. Μας ε, επιβεβαιώσατε με ένα τρόπο ο οποίος είναι πραγματικά τρομερός, τρομακτικός, το, την έκταση του προβλήματος με τις πληροφορίες αυτές που μας φέρετε. Είναι σαν να βρισκόμαστε στο 1914, ενώ είμαστε στον 21ο αιώνα. Είναι μια άσκηση πολιτικής που δεν θέλαμε να την ξαναδούμε. Ο κύριος Πούτιν, ο πρώην επικεφαλής της ΚΑΓΕΜΠΕ, όταν λέει αυτά τα οποία λέει δεν προκαλεί καμία εμπιστοσύνη σε εμά τους Γερμανούς οι οποίοι έχουμε γνωρίσει το παρελθόν αυτό. Βλέπουμε να είναι απλώς μια νέα μορφή υπεριαλισμού. ένας τρόπος να ενσωματώσει την Ουκρανία στη σφαίρα επιρροής της ε, Ρωσίας σαν μια παλιά Σοβιετική Ένωση. Εδώ πέρα όμω βλέπουμε ότι έχουν πέσει οι μάσκες και είναι σαφείς οι προθέσει του. Προφανώς είναι σημαντικό να δώσουμε την αλληλεγγύη μας και την υποστήριξή μας, αλλά πιστεύω ότι μια συμφωνία σύνδεση αυτή τη στιγμή δεν πρόκειται να βοηθήσει σε τίποτα. Δεν θα πετύχει αυτά που θέλαν οι διαδηλωτέ στην πλατεία Μαϊντάν. Κάτι το οποίο είναι πιο σημαντικό είναι ένα σχέδιο δράσης για την ένταξη της Ουκρανίας που είχε ε, αποφασιστεί το 2008 στο Βουκουρέστι και με ελαφρά την καρδία ουσιαστικά δεν εφαρμόστηκε. Ξέρω ότι οι βαλτικές χώρες ήταν, ε, για αυτές ήταν πιο σημαντικό να είναι τμήμα του ΝΑΤΟ και όχι της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε πρώτη προτεραιότητα, γιατί προφανώς η εδαφική ακαιρεότητα είναι πολύ πιο σημαντική. Αλλά όταν βλέπουμε την ε, στάση του Μετβέντεφ και του Πούτιν και το δόγμα αυτό ότι η Ρωσία θα πρέπει να επέμβει όπου βρίσκονται Ρώσοι πολίτες, βλέπουμε ότι αυτή η μέθοδος είναι ακριβώς η ίδια που χρησιμοποιήθηκε για την εισβολή στο, στην Πράγα το 1968 ή το 1980 στο Αφγανιστάν. Είναι τρομερό αυτό το πράγμα που συμβαίνει. Τάνοκ. Αγαπητέ Μπόρι, σε καλωσορίζω εξ ονόματος της ομάδας των συντηρητικών και δημοκρατών. Σε υποδεχόμαστε εδώ σαν εκπρόσωπο μιας νέας δημοκρατικής Ουκρανίας με ένα δυτικού τύπου θα έλεγα δημοκρατικό μέλλον. Δυστυχώς βλέπουμε τώρα ότι παραβιάζεται η διεθνής τάξη από τη ρωσική ε, ε, ομοσπονδία υπό τη δικτατορία θα έλεγε κανείς πλέον του Πουτίν ο οποίος τα κάνει όλα μόνος του σχετικά με το κείμενο εγγύσεων το μνημόνιο της Βουδαπέστης οι Αμερικανοί λέει ότι είναι κάποιες διαβεβαιώσεις αλλά οι μόνες κυρώσεις είναι περνούν μέσα από διαβουλεύσεις τι ακριβώς περιμένετε εσείς από την εφαρμογή τους από ό,τι μου φαίνεται και παρακολουθώ τα θέματα αυτά και διάβασα και κάτι σήμερα, στην ουσία ε, ακούστηκαν πάρα πολλά ψέματα. Ο Πουτίν και η Κάγκεμπέ ε, οργανώνουν την προσπάθεια αυτή εδώ και πάρα πολύ καιρό λένε ότι 600.000 ρωσόφωνοι από την Ουκρανία αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τη χώρα και να ζητήσουν προστασία στην Ρωσία αλλά από την άλλη ξέρουμε ότι και διάφοροι αλητήριοι στην υπηρεσία των υπηρεσιών των μυστικών προκάλεσαν πάρα πολλά επεισόδια αιματηρά μάλιστα σε πόλεις όπως το Ντονέτσκ. Όπως είπε ο Τσόρτσιλ, τον πόλεμο δεν τον θέλουμε ποτέ. Από την άλλη δεν ξέρω αν οι κυρώσεις όπως ε, αυτές που επιβάλαμε στους Ιρανούς Επίσης θα πρέπει να δείξει την ε, αλληλεγγύη της με την Ουκρανία και η Τουρκία και ε, ε, επίσης και με τους Τατάρους οι οποίοι έχουν υποφέρει φρικτά από το Στάλιν και από τους Ρώσους ήδη από τη δεκαετία του 30. Όλα αυτά θυμίζουν το τι συνέβη στη δεκαετία του 60 στην Τσεχοσλοβακία, τα λέω όλα αυτά μαζί και το θέμα τώρα του δημοψηφίσματος στην Κρυμαία έτσι και αλλιώ αυτό δεν είναι κάτι το οποίο θα μπορούσε να επιτρέψει ποτέ στη Ρωσία να γίνει ο Πουτίν. Εκ μέρους του ΑΚΕΛ και της Γκουε θα ήθελα να εκφράσω τη συμπαράστασή μας στον Ουκρανικό λαό την πίστη μας ότι έχει δικαίωμα στο μέλλον του και μόνον αυτός δικαιούται να αποφασίσει για το μέλλον του. Ε, θέλω επίσης να πω όμως, και ας μου επιτραπεί αυτό, ότι βρίσκω αυτή τη συζήτηση λίγο μονοπλευρή. Ε, όχι γιατί ε, εκφράζονται απόψεις μόνο από μια απόψη από τους συναδέλφους. Αυτό, αυτό είναι δικαίωμα και υποχρέωση. Αλλά δεν μπορώ να καταλάβω γιατί στο πάνελ ε, η διαφορετική άποψη απουσιάζει. Υπάρχει μια μόνο αλήθεια για αυτό το ζήτημα. Εγώ θεωρώ ότι δεν μπορεί να υπάρξει μια ουσιαστική συζήτηση αν δεν ακούσω και μια διαφορετική άποψη πάνω σε αυτό το ζήτημα, η οποία υπάρχει. Και διαρωτούμε πού χάθηκε η realpolitik πολλών ανθρώπων σε αυτή την αίθουσα, την οποία υπερασπίζονται σε άλλες περιπτώσεις και τώρα αγνοούν πλήρως την, την ανάγκη η, η πραγματικότητα να ορίσει τη συμπεριφορά μας έτσι ώστε να μην επέλθουν περισσότερα δεινά στον Ουκρανικό λαό. Ε, με αυτά τα δεδομένα είναι που υποστηρίζω ότι πρέπει και η Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει την ίδια συγκράτηση απέναντι σε αυτό το ζήτημα όπως την συγκράτηση που απαιτεί από άλλους. Uh, Πρώτα απ' όλα, αγαπητοί φίλοι, θέλω να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου σε εσά για το ενδιαφέρον σας, για το σαφές ενδιαφέρον που φάνηκε από τις δηλώσεις σας και από τα ερωτήματά σας. Για να απαντήσω στα πρώτα ερωτήματα που έθεσε ο Ιγνάσιος Αλαφράνκα, θέλω να πω ότι πράγματι πιστεύω ότι οι οικονομικές κυρώσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της Ρωσίας θα είναι ένα είδος κρύου ντους για τη Ρωσία. Οι οικονομικές κυρώσεις με την ευρύτερη έννοια, όχι μονάχα δηλαδή κυρώσεις εναντίον αξιωματούχων της Ρωσίας, που είναι αυτοί οι οποίοι πήραν την απόφαση για την επίθεση κατά της Ουκρανίας. Για το ΝΑΤΟ, αγαπητοί συνάδελφοι, εμείς ως Ουκρανοί καταλαβαίνουμε ότι εμείς και μόνο εμείς θα πρέπει να εξασφαλίσουμε την άμυνα της χώρας μας. Συγχρόνως, το ΝΑΤΟ είναι ένα πολύ σημαντικό όργανο παγκόσμιας ασφάλειας. Έχει παίξει και παίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο για την ασφάλεια της Ευρώπης και την ευρύτερη ασφάλεια στην περιοχή της Ευρώπης και του Ατλαντικού. Θέλω να σας υπενθυμίσω σχετικά ότι η Ουκρανία το 2006 υπέβαλε μια αίτηση για να γίνει μέλος της ε, συμμαχίας του ΝΑΤΟ. Το 2008, στην διάσκεψη κορυφής του ΝΑΤΟ στο Βουκουρέστι, η απάντηση ήταν ότι η διάσκεψη κορυφής, κορυφής καλωσορίζει τις προσδοκίες του, της Ουκρανίας για να γίνει μέλος του ΝΑΤΟ και συμφώνησε ότι θα γίνει εν καιρό μέλος του ΝΑΤΟ η Ουκρανία. Και εγώ απλώς σας υπενθυμίζω την απόφαση του Βουκουρεστίου στις 3 Απριλίου 2008. Τι θα γίνεται τώρα όμως. Εγώ ήμουνα, είμαι και θα είμαι πάντα ιδιαίτερα στεναρός υπέρμαχος της ιδέας του να γίνει η Ουκρανία μέλος και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ. Συγχρόνως όμως θα πρέπει να σας πω ότι αυτή τη στιγμή στο Ουκρανικό Κοινοβούλιο δεν μπορούμε να αποκλείσουμε μια κίνηση για ένταξη στο ΝΑΤΟ. Εγώ δεν μπορώ να αποκλείσω να γίνει κάποια τέτοια πρόταση. Και ξέρω ότι ένα τέτοιο αντίστοιχο ψήφισμα, σχέδιο ψηφίσματος, είχε υποβληθεί, έχει υποβληθεί στο Ουκρανικό Κοινοβούλιο και μπορεί να τύχει ψηφοφορία αύριο. Εάν πράγματι τεθεί σε ψηφοφορία αυτό το σχέδιο, εγώ πιστεύω ότι είναι πολύ πιθανό να εγκριθεί από την πλειοψηφία των μελών του Κοινοβουλίου μας. Για την Κρυμαία, σε ποιον θα πρέπει να απευθυνθούμε. Αυτό που έγινε στην Κρυμαία πριν οι Ρώσοι με ανοιχτό τρόπο εισέβαλαν στην Κρυμαία. Καταρχήν προετοίμασαν πολιτικά την κατάσταση χρησιμοποιώντας τους συμμάχους τους στο Κοινοβούλιο της Κρυμαίας και την κυβέρνηση της Κρυμαίας με ένα τρόπο ο οποίος ήταν παράνομος, με παράνομες μεθόδους, ε, ανέτρεψαν την κυβέρνηση της Κρυμαίας, γιατί δεν είχαν επαρκή πλειοψηφία μεταξύ αυτών που πήραν αυτή την απόφαση. Η απόφαση αυτή για μας δεν έχει νομιμότητα. Και οι Ρώσοι έχουν επιβάλει στην Κρυμαία ως ηγέτη κάποιον ο οποίος είναι γνωστός ως επικεφαλής εγκληματικών συμμοριών στην Κρυμαία, τον κύριο Αξόνοφ, ο, ο οποίος τώρα αυτός είναι ο, ο επικεφαλής της κυβέρνησης της Κρυμαίας με ακολουθώντας τις εντολές των Ρώσων. Να μιλήσουμε μαζί του. Δεν έχει κανένα νόημα αυτό. Ο ασκόντη προεδρία στην ε, Ουκρανία έχει ε, διορίσει τον κύριο Κουνίτσιν ως εκπρόσωπό του στην Κρυμαία. Είναι ένας γνωστός πολιτικός Κρυμαίας. Η κατάσταση όμως επισκιάζεται απόλυτα από την παρουσία των Ρώσων. Οι Ρώσοι με τους ε, συμμάχους τους και τους αντιπροσώπους τους ασκούν την εξουσία και φυσικά έχουν και τη στρατιωτική δύναμη στην Κρυμαία. Για τα δικαιώματα των εθνοτικών μειονοτήτων. Αν θέλετε το πιστέψετε ή όχι. Αλλά οι Τατάροι της Κρυμαίας, μεταξύ όλων αυτών των εθνοτικών ομάδων στην Κρυμαία, είναι αυτοί οι οποίοι υποστηρίζουν περισσότερο την Ουκρανία, την Ουκρανική θέση στην Κρυμαία. Και παρά τις προσπάθειες που έχουν καταβληθεί για να δημιουργηθεί κάποιο μίσος μετά των Τατάρων της Κρυμαίας και του υπόλοιπου πληθυσμού της Κρυμαίας, οι Τάταροι έχουν καταφέρει να συμφωνήσουν με τους εκπροσώπους των βετεράνων του Αφγανιστάν, αυτών δηλαδή που πολέμησαν στην εκστρατεία του Αφγανιστάν με τη Σοβιετική Ένωση, οπότε και πάλι εξακολουθούν να ε, περιπολούν στις πόλεις της Συμφερόπολης και να εξασφαλίσουν την τάξη. Οι Τατάροι μαζί με τους βετεράνους του Αφγανιστάν. Η υπογραφή της συμφωνίας σύνδεσης. Εγώ δεν ξέρω πώς μια τέτοια συμφωνία η οποία είχε τύχει διαπραγματεύσεων για πάρα πολλά χρόνια, από το 2007 μέχρι τώρα, πώς μια τέτοια συμφωνία αν υπογραφεί αυτό θα οδηγήσει σε τάσεις, σε εντάσεις. Γιατί ξεκινήσαν οι διαμαρτυρίες στην πλατεία Μαϊντάν. Γιατί ο λαός δεν συμφωνούσε με τις αρχές της χώρας του που αποφάσισαν την τελευταία στιγμή να μην υπογράψουν αυτήν την συμφωνία σύνδεση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είμαι βέβαιος λοιπόν ότι η πλειοψηφία του Κοινοβουλίου πάνω από 300 δηλαδή βουλευτές, θα υποστηρίξουν και υποστηρίζουν πράγματι την υπογραφή της Συμφωνίας Σύνδεσης. Και αυτή η συνταγματική πλειοψηφία εκπροσωπεί και την πλειοψηφία των Ουκρανών. Πιστεύω λοιπόν ότι ο λαός υποστηρίζει απερίφραστα την έγκριση της Συμφωνίας Σύνδεσης. Για τις εγγύησεις τώρα και τις διασφαλίσεις. Όταν βρέθηκα στο μέσο των διαπραγματεύσεων αυτών για το μνημόνιο της Βουδαπέστης, εγώ θυμάμαι πολύ καλά, ότι μια χώρα η οποία είναι από την άλλη πλευρά του ωκεανού επέμεινε να μην χρησιμοποιηθεί η διατύπωση εγγυήσεις αλλά διαβεβαιώσεις. Εγώ καταλαβαίνω ποια είναι διαφορά και εσείς καταλαβαίνετε ποια είναι διαφορά μεταξύ διαβεβαιώσεων και εγγύησεων. Αλλά σε όλες τις άλλες γλώσσες δεν υπάρχει καμία διαφορετική ερμηνεία από τη λέξη εγγύηση. Αυτό ισχύει στα ρώσικα, ισχύει στα ουκρανικά, αν δεν κάνω λάθος και στα γερμανικά η μετάφραση για τις ε, διαβεβαιώσεις αυτές σε στα αγγλικά μεταφράστηκε ως εγγύησης. Επομένως προσδοκούμε ότι οι εγγύητρες χώρες που μας έδωσαν αυτές τις διαβεβαιώσεις ασφαλείας θα εφαρμόσουν αυτές τις εγγύησεις, θα τηρήσουν το καθήκον τους και θα σταματήσουν την ε, εισβολή, την επίθεση που γίνεται από μια χώρα που είναι και αυτή εγγύητρια του Μνημονίου της Βουδαπέστης. Ποιες είναι δυνατότητες για κυρώσεις. Κατά τη δική μου άποψη, όλα μπορούν να γίνουν εκτός από τη χρήση της ε, βίας, από μια στρατιωτική ε, επέμβαση. Όλα αυτά λοιπόν θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν εναντίον τη Ρωσία και αυτό συμπεριλαμβάνει τι οικονομικέ κυρώσει. Νομίζω ότι έχουμε μεγάλο περιθώριο να χρησιμοποιήσουμε οικονομικέ κυρώσει εναντίον τη Ρωσία. Τώρα, το αν έχει νόημα αυτή τη στιγμή να υπογραφεί η Συμφωνία Σύνδεση, όπω είπα και προηγουμένω, νομίζω θα βοηθήσει πολύ. Θα βοηθήσει και τα εκατομμύρια των Ουκρανών που ειρηνικά διαδήλωσαν για ένα ευρωπαϊκό μέλλον της Ουκρανίας. Θα είναι μια μορφή ανταμοιβή για τον αγώνα τους. Και επίσης το να τους δοθεί ένα καθεστώς μη υποχρέωσης προξενικής βίζας για να ταξιδεύουν στην Ευρώπη. Αυτό περιμένουν λοιπόν εκατομμύρια Ουκρανών από εσά. Και φυσικά την προοπτική να ενταχθεί η Ουκρανία πλήρως στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι κάτι το οποίο συζητάτε ήδη αυτές τις τελευταίες μέρες στα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πολύ σωστά. Οι κυρώσει λοιπόν μπορεί να μην είναι εναντίον της ε, χώρας ε, η οποία έχει εισβάλει στην Ουκρανία αλλά και εναντίον των αξιωματούχων αυτής της χώρας. Και συμφωνώ μαζί σου Τσάρλς ότι το δημοψήφισμα στην Κρυμαία που αντιτίθεται με τις ρήτρες του κρημαϊκού συντάγματος δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι έχει νόμιμο χαρακτήρα. Από την αρχή. Εμείς έχουμε τονίσει ότι δεν μπορεί να είναι αποδεκτό το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος αυτού γιατί ήδη από την αρχή είναι παράνομο. σχετικά με την τελευταία άποψη σε σχέση με το ότι εκφράζω μία μονομερή θέση. Κοιτάξτε, εγώ εκπροσωπώ τις απόψεις του Ουκρανικού λαού που εκφράστηκε στο Μαϊντάν τις τρεις τελευταίες εβδομάδες. Πάνω από 300 μέλη του Κοινοβουλίου υπερψήφισαν α, τα, τις απόψεις που έχω τώρα για τα θέματα τα οποία συζητάμε δηλαδή πάνω από την απαιτούμενη συνταγματική πλειοψηφία υποστήριξαν την νέα Ουκρανική κυβέρνηση. Συνεπώς δεν εκφράζω μόνο μερίς απόψεις. Εγώ εκφράζω τις απόψεις των, της κυβέρνησης η οποία υποστηρίζεται και από τους τέους αντιπάλους. Λοιπόν, ε, έχουμε να κάνουμε με μια κυβέρνηση προϊόν της δημοκρατικής επανάστασης που συνέβη τις τελευταίες μέρες στην Ουκρανία. Σας ευχαριστώ για όλα. Everyone has one minute. First, Mr. Thank you, Chairman. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Γνωριζόμαστε εδώ και αρκετά χρόνια. Θα ήθελα να επαναλάβω αυτό που είχα πει σε με άλλη αφορμή τον μήνα Σεπτέμβριο του προηγούμενου χρόνου ότι θα πρέπει εμείς να προτείνουμε να πάρει το Νόμπελ ο Πουτίν για την γιατί είναι πολύ καλός οφθαλμίατρος από ό,τι φαίνεται και στην ουσία μας κάνει να βλέπουμε και εμάς τη Ρωσία με διαφορετικό τρόπο. Εν πάση περιπτώσει, ε, εσύ γνωρίζεις τον Πούτιν καλύτερα από μένα. Τι θέλει ο Πούτιν, θέλει την Κρυμαία όπως λέγουν ορισμένοι αμπειρογνώμονες. Θέλει το ανατολικό τμήμα της Ουκρανίας, θέλει όλη την Ουκρανία. Τι θέλει, εν πάση περιπτώσει, ο Πουτίν. Δεύτερη ερώτηση, τι μπορούμε εμείς σαν Ευρωπαίοι να κάνουμε έτσι ώστε να μην το πετύχει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν μας μιλήσατε ακόμα καθόλου για τη συνεργασία μεταξύ του ΟΣΑ και του ΟΗΕ στο βαθμό που θα μπορούσαν να συμμετέχουν και αυτοί σε ό,τι αφορά δηλαδή την εξέβρεση μιας διπλωματικής οδού. Και τι θα γίνει αν αύριο ή μεθαύριο οι G7 συναντηθούν γιατί θεωρώ ότι δεν θα υπάρξει λύση χωρίς τη Ρωσία ακόμα και αν ε, ο Πούτιν ε, Ανακηρυχτεί τρελός ή βάση περιπτώσει. Δεν πιστεύω ότι έχει νόημα να μιλάμε σήμερα για κυρώσεις, γιατί ένα μεγάλο τμήμα του ρουσικού πληθυσμού θα ε, έκανε ένα μποϊκοτάρισμα. Νομίζω ότι ο μοναδικός τρόπος λοιπόν είναι μια διπλωματική οδός. Και σε ό,τι αφορά την υπογραφή της Συμφωνίας Σύνδεσης και για τον ΝΑΤΟ, θεωρώ ότι αυτό θα ήταν μια ε, ένα δούμε προς τα πίσω. Σας ευχαριστώ κύριε Τρασιούκ. Εγώ είμαι από την Κροατία και βλέπω ότι υπάρχουν πολλές ομοιότητες μεταξύ των χαρακτηριστικών του Πούτιν ε, σήμερα και του Σλόμποντα Μιλόσεβιτ στην δεκαετία του 90. Δεν είναι οι ίδιε οι καταστάσει φυσικά, αλλά υπάρχουν πολλές ομοιότητες και θα ήθελα να τονίσω το εξής. Εγώ βλέπω και ομοιότητες σε ό,τι αφορά την ε, κατανομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε ό,τι αφορά του, τη διεθνή κοινότητα και τους στόχους που επιδιώκει ο καθένας. Είναι σημαντικό να δείξουμε αλληλεγγύη και μάλιστα με συγκεκριμένα μέτρα. Ήσασταν πάρα πολύ ακριβείς και πιστεύω ότι θα πρέπει σήμερα να φύγουμε από τη σημερινή συνεδρίαση με ένα σαφές μήνυμα. Το μήνυμα της, ε, των σαφών μέτρων αλληλεγγύης από πλευρά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ο Σερ Ρόμπερτ. Να υποστηρίξω και εγώ την υποστήριξή μου στην προσπάθειά σας. Προφανώς ε, τα μέσα ενημέρωση στα ρωσικά λέγουν ότι ε, ένας άμεσα δημοκρατικά εκλεγμένος πρόεδρος ε, διώχθηκε. Δεύτερον λένε ότι υπάρχει μια συμφωνία για την υποστήριξη του στόλου της Μαύρης Θάλασσας και εξέφρασαν αμφιβολίες για την ασφάλεια του στόλου τους. Γιατί δεν ακούστηκε από πλευρά σας μια ξεκάθαρη ε, θέση για το τι θα γίνει με τον ρωσικό στόλο μετά το 2017. Και βλέπω εδώ ότι η Κίνα υποστηρίζει, είπε σήμερα, την ρωσική θέση. Τι σημαίνει αυτό. Ε, εκτός από το ότι βέβαια το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών δεν έχει πλέον κανένα ρόλο να παίξει. Η κυρία Λιούψεβα έχει ζητήσει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ομιλώ τη Βουλγαρική. Αγαπητέ κύριε Τάρασουκ, ε, είμαστε όλοι μάρτυρες σήμερα μιας συνεχούς κλιμάκωσης της ε, κρίσιμης κατάστασης στη χώρα σας παρά τις προσπάθειες τις οποίες έχουμε κάνει σαν Ευρωπαϊκή Ένωση και εμείς και άλλοι βέβαια. Είναι όμως σαφές ότι πρέπει να εκφραστούμε με ομόφωνη άποψη. Είμαστε όλοι φίλοι του Ουκρανικού λαού και όλοι πρέπει να είμαστε αλληλέγγυοι με τον Ουκρανικό λαό και την αλληλεγγύη μας αυτή θα πρέπει να την επιδείξουμε με συγκεκριμένο τρόπο να εγγυηθούμε την εξέβρεση ειρηνικής λύσης και να διασφαλίσουμε την ειρήνη και την ακαιρεότητα της Ουκρανίας γνωρίζετε ότι δεν θα πρέπει να υπάρχουν απειλές για τις μειονότητες. Και εδώ έρχεται μία ερώτηση από πλευράς μου. Ο νόμος, ο σχετικός ε, με την ε, ελευθερία χρήσης των μειονοτικών γλωσσών είναι ένας καλός νόμος Από την άλλη το θέμα των κυρώσεων είναι κάτι το οποίο μπορεί να συζητηθεί αλλά δεν θα πρέπει να φύγει τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και τους πολίτες της χώρας αυτής. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε, σας ευχαριστώ κύριε Ταρασούκ που ήρθατε εδώ για να μας ε, παρουσιάσετε τη θέση σας. Θα ήθελα εξ αρχής να πω ότι είμαστε αλληλέγγυοι και υποστηρίζουμε την αλληλεγγύη προς την κυβέρνηση στο Κίεβο. Είμαστε ενώπιον μιας μεγάλης πρόκλησης και νομίζω ότι η διεθνής κοινότητα θα πρέπει να καταβάλει μεγάλες προσπάθειες και θα πρέπει να φροντίσει να αποκλιμακωθεί η κατάσταση. Είχα τηλεφωνική επαφή σήμερα με φίλους από την Κρυμαία. Η κατάσταση είναι πάρα πολύ σοβαρή. Ο ψυχολογικός πόλεμος, ε, ο φόβος που επικρατεί μεταξύ του κόσμου, η παρουσία ε, των στρατευμάτων στον κόσμο, κανείς που δεν μπορεί να φύγει, κανείς δεν μπορεί να φύγει από την Χερσόνησο. Όλα αυτά λοιπόν δεν θα πρέπει να υπάρξουν περαιτέρω προκλήσεις γιατί σε την περίπτωση αυτή θα ήταν έντονη η κλιμάκωση. Μία ερώτηση σε ό,τι αφορά και τον κύριο Άτκινς η Ρώσοι ασφαλώς έχουν διάφορες δικαιολογίε που προβάλλουν σε ό,τι αφορά και την σεβαστό πολύ. Το Κίεβο αυτή, αυτό το μήνυμα θέλει να αποστείλει. Eh, ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ τον κύριο Τασιόπ για την παρουσία του πέραν της καταδίκης ρωσικής ε, επέμβασης θέλω να κάνω και κάποια ερωτήματα για να μπορέσουμε με τον τρόπο αυτό να έχουμε μια πιο σαφή εικόνα της κατάστασης. Θεωρείτε όπως ζητεί ο αρχηγός της ομάδας μου και ζητούν διάφοροι διπλωματικοί κύκλοι θεωρείτε ότι πρέπει να συμπεριλάβουμε και τη Ρωσία στον πολιτικό διάλογο γιατί η απομόνωση της Ρωσίας παίζει κάποιο ρόλο στη δυναμική των πραγμάτων. Η Ρωσία είναι μια μεγάλη δύναμη και δεν πρέπει να βρεθεί σε ένα αδιέξοδο γιατί αυτό μπορεί να οδηγήσει σε μια μεγαλύτερη κλιμάκωση της βίας. Και για την Ουκρανία. <clears throat> Θεωρείται ότι η Ουκρανία θα πρέπει να επαναφέρει την νομοθεσία που προστατεύει τις μειονότητες, τις ε, γλωσσικές μειονότητες, μεταξύ άλλων και, τον, και τη ρωσόφωνη μειονότητα. Και τι γίνεται με τις των ρωσόφιλων Ουκρανών πολιτών στην ε, ε, ανατολική περιοχή της Ουκρανίας και την Κρυμαία και αυτός και η στάση του κυρίου Μπερεζίνσκι του Ναβάρχου του στόλου της Κρυμαίας ο οποίος έχει πει ότι θα ακολουθήσει τις αποφάσεις της κυβέρνησης Κρυμαίας εκεί. Ο κύριος Βούλιανιτς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε είναι αρκετά σαφέ τι έγινε στην Ουκρανία. Όλοι το καταλαβαίνουν και το ξέρουν. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Ταρασίου που μας έδωσε την πλήρη εικόνα της κατάστασης. Από την άλλη πλευρά, η Ρωσία δεν δίνει και μεγάλη σημασία στα δημοκρατικά δικαιώματα, τα ανθρώπινα δικαιώματα κτλ. Μια τέτοια δικτατορία σέβεται μονάχα το δικό της εθνικό συμφέρον. Έχει πάρει λοιπόν τα απαραίτητα μέτρα για να προστατεύσει το εθνικό συμφέρον όπως το αντιλαμβάνονται ήδη. Δεν θα αλλάξουμε τη Ρωσία. Δεν έχουμε τη δύναμη, δεν έχουμε καν τη θέληση να το κάνουμε. Μπορούμε όμως να βοηθήσουμε την Ουκρανία. Αλλά πρέπει να είμαστε σε θέση να καταλάβουμε τι τίμημα θα έχει αυτή η βοήθεια. Δεν μπορούμε να βοηθήσουμε σε στρατιωτικό επίπεδο. Μπορούμε να βοηθήσουμε πολιτικά μας, μπορούμε να βοηθήσουμε πάρα πολύ και μπορούμε να βοηθήσουμε την Ουκρανία οικονομικά, στο οικονομικό επίπεδο. Με την προϋπόθεση ότι τα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι έτοιμα να το κάνουν. Τα έχετε ρωτήσει αν αυτή είναι η θέλησή τους ή όχι. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ λέει και ο Πρόεδρος. Ο κύριος Ταρασούκ για να απαντήσει. Για μια ακόμη φορά θα ήθελα να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου για τις πολύ καλές και ενδιαφέρουσες ερωτήσεις σας και για το ενδιαφέρον γενικά το οποίο επιδεικνύεται. Κάποιοι από εσά ρώτησαν τι θέλει ο Πουτίν. Θέλει να ελέγξει την Κρυμαία μόνο, θέλει να ελέγξει την Ανατολική Ουκρανία ή θέλει να ελέγξει το σύνολο της Ουκρανίας. Εγώ εδώ μπορώ να απαντήσω στην ερώτησή σας σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες. Από ό,τι βλέπω οι Ρώσοι έχουν συγκεντρώσει στρατεύματα στα ανατολικά μας σύνορα, Χάρκοβο, Λογάνσκα και Ντονιέτσκα, στους τρεις νομούς, τα τρία όμπλαστα αυτής της περιοχής. Λοιπόν, ε, εγώ ασχολούμαι με τους Ρώσους και έχουμε να αντιμετωπίσουμε τους Ρώσους από τότε που ήμασταν τμήματα όλοι της Σοβιετικής Ένωσης και μπορώ να πω το εξής. Οι Ρώσοι ποτέ δεν θα είναι ικανοποιημένοι με μία μικρή παραχώρηση όσο σημαντική και αν είναι από την Ουκρανία. Η μόνη παραχώρηση με την οποία θα ικανοποιηθούν είναι να ελέγξουν το σύνολο της χώρας. Αυτή είναι η μοναδική για τους Ρώσους ε, επιδιωκόμενη λύση. Να πω επίσης ότι ανάμεσα στις τέως Σοβιετικές Δημοκρατίες μόνο η Ουκρανία είχε αντισταθεί θα έλεγα όλα αυτά τα χρόνια ε, στον ρωσικό έλεγχο και η Ουκρανία ήταν αυτή η οποία είχε ασκήσει τη δική της εξωτερική πολιτική σε σχέση με άλλες Σοβιετικές Δημοκρατίες. How Πώς μπορούμε να σταματήσουμε τον Πουτίν με δύο τρόπους. Πρώτον ο ίδιος του ο λαός θα τον σταματήσει κάποια στιγμή. Και δεύτερον μέσω της πίεσης της διεθνούς κοινότητας αυτό βέβαια θα εξαρτηθεί από το πόσο σοβαρή θα είναι αναλαμβάνοντας τις ευθύνες της η διεθνής κοινότητα. Σχετικά με τον ΟΑΣΕ Φυσικά και εμείς ε, ε, προσδοκούμε από την παρέμβαση του ΟΑΣΕ σαν μέσο διεθνού συνεργασίας. Από την άλλη ο ΟΑΣΕ εξαρτάται φυσικά και αυτός από τις απόψεις των Ρώσων και γι' αυτό δεν είμαστε πάρα πολύ αισιόδοξοι. Η δημοπλατεία πρέπει να είναι ε, πρώτη και δραστήρια αλλά οι Ρώσοι από ό,τι φαίνεται δεν ε, ε, συμφωνούν με αυτή την άποψη και αποφάσισαν χωρίς διπλωματικές συζητήσεις να εισβάλλουν σε ένα τμήμα της ε, Ουκρανίας. Και οι Ρώσοι είπατε ότι μπορεί να βλάπτουν τους πολίτες. Να θέσω το ερώτημα με διαφορετικό τρόπο. Το τίμημα που πληρώνουν οι Ρώσοι για την εισβολή της Ουκρανίας είναι αρκετά υψηλό νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο θα επηρεάσει το σύνολο των Ρώσων γιατί είναι χρήματα τα οποία τα παίρνουν από κοινωνικά προγράμματα και τα οποία θα έπρεπε να ωφελήσουν τους Ρώσους πολίτες. Αλλιώς τα χρήματα αυτά θα χανόντουσαν, θα χαθούν μάλλον ακριβώς την προσπάθεια αυτή της στρατιωτικής εισβολής για τον Σερ Ρόμπερτ. Μιλήσατε για την ανατροπή του δημοκρατικά νόμιμα εκλεγμένου Προέδρου της Ουκρανίας. Κοιτάξτε, ε, πολλοί δεν αμφισβητούν το ότι ο Γιαννούκοβιτς εξελέγει με δημοκρατικό τρόπο, αλλά κάποιοι πάλι από την άλλη στην Ουκρανία το πιστεύουν αυτό. Αλλά εμείς στην περίπτωση αυτή δεν συζητάμε για την ανατροπή του Προέδρου της Ουκρανίας εμείς μιλάμε για έναν πρόεδρο της χώρας ο οποίος διέφυγε με ανεύθυνο τρόπο από μόνος του και δεν εφάρμοσε ε, ενέργειες ε, οι οποίες, ε, τις οποίες ο ίδιος είχε αναλάβει να εφαρμόσει και έβαλε την υπογραφή του γι' αυτό στις 21 Φεβρουαρίου και ο Μπρόκ ήταν παρόν όταν υπεγράφει η συμφωνία με τον Γιαννούκοβιτς σκοπιμότατα σε εισαγωγικά λοιπόν έφυγε από τη χώρα και δεν εφάρμοσε τη συμφωνία στην οποία είχε συνυπογράψει, δεν είχε εφαρμόσει τις αλλαγές τις συνταγματικές τις οποίες ανέλαβε την υποχρέωση μετά από ψήφο του Κοινοβουλίου να εφαρμόσει. Προτίμησε να διαφύγει στο εξωτερικό. Έχουμε την αίσθηση λοιπόν ότι το πρόσωπο αυτό διέπραξε κάτι το οποίο ε, στην ουσία ισοδυναμεί με προδοσία. Αφού υπέγραψε τη συμφωνία αυτή, ε, εγώ κατέθεσα στο Κοινοβούλιο την πρόταση ψηφίσματος λέγοντας ότι η συμφωνία του Χάρκιβ στην ουσία ε, επέβαλε την παρουσία των ναυτικών ρωσικών δυνάμεων στο έδαφος μας μέχρι το 2042 και αυτό ισοδυναμεί με εθνική προδοσία. Δεν υπήρχε έτσι κι αλλιώς η δυνατότητα συνταγματικά ούτε καν μέχρι το 2017 γιατί η συμφωνία η οποία ε, υπάρχει δεν μπορεί να ξεπεράσει το 2017 με οδήποτε τρόπο χρονικά. Νομίζω λοιπόν ότι η μεγάλη πλειοψηφία της Ουκρανικής Βουλής καταγγέλει τη συμφωνία αυτή του Χάρκοφ που δίνει την δυνατότητα στους Ρώσους να παραμείνουν έστω και μέχρι το 2017. Τώρα για την Κίνα. Εγώ δεν γνωρίζω κάποιο γεγονός το οποίο να ερμηνεύεται ε, με υποστήριξη της Ρωσίας από την Κίνα. Ε, στο Συμβούλιο Ασφαλείας οι Κινέζοι είπαν <coughs> ότι είναι και πάντα θα είναι ε, αυτοί που θα σέβονται την εδαφική ακαιρεότητα ασδήποτε χώρας. Για τις εθνικές μειονότητες γίνονται σεβαστές. Και αυτό το είπε και ο Επίτροπος του Ισοασέ ε, για τις εθνικές μειονότητες. Καλέστε τον στη συνεδρίαση της Επιτροπής σας και ρωτήστε την άποψή του να σας πει πώς αξιολογεί τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ουκρανία. Σχετικά τώρα με τον περίφημο νόμο για τη γλωσσική ελευθερία ή την ελευθερία χρήσης μειονοτικών γλωσσών, ο νόμος ο οποίος ψηφίστηκε πρόσφατα κατά της χρήσης της γλώσσας αυτής κατετέθη από πολιτικούς αντιπάλους. Ήταν ένας νόμος ο οποίος φρόντιζε αποκλειστικά τους Ρώσους εις βάρος την ρωσική μειονότητα δηλαδή, εις βάρος όλων των άλλων μειονοτήτων της Ουκρανίας μεταξύ των οποίων και των ίδιων των Ουκρανών. Υπήρξε μια πολιτική συμφωνία κάποια στιγμή έτσι και αλλιώ ο Προεδρεύων δεν είχε υπογράψει ε, τον νόμο τον καινούριο, δεν έχει εφαρμοστεί ακόμα και αποφασίστηκε οι πολιτικές ομάδες στην Ουκρανική Βουλή να συνέλθουν και να καταθέσουν μια νέα πρόταση νόμου σχετικά με την προστασία των εθνικών μειονοτήτων και των μειονοτικών τους γλωσσών. Να σας πω εδώ ότι η Ουκρανία έχει προσυπογράψει και την χάρτα του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των γλωσσικών ε, μειονοτικών δικαιωμάτων. <coughs> Και σεβόμαστε πλήρως αυτά τα οποία προβλέπει αυτή η συμφωνία για τις ε, μειονοτικές γλώσσες. Σας ευχαριστώ και πάλι λοιπόν για τα αισθήματα αλληλεγγύης που εκφράσατε. Ευχαριστώ πολύ. Λέω πρόεδρος Μπροκ. Πιστεύω ότι ήταν πάρα πολύ σημαντικές όλες αυτές οι πληροφορίες και διευκρινήσεις που πήραμε από τον κύριο Θάσιονου. Και στις, ε, 3.30, θα, στις 4.30 συγγνώμη, ο θα μας πληροφορήσει για τις συζητήσεις του Συμβουλίου Υπουργών Εξωτερικών. Ίσως είναι σημαντικό να μείνετε και για αυτή την ενημέρωση. Αγαπητέ Μπάρις, ευχαριστώ πάρα πολύ για τον κόπο που έκανες να έρθεις εδώ και μπορείς να είσαι σίγουρος ότι η μεγάλη πλειοψηφία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι έτοιμη να εκφράσει την ε, αλληλεγγύη της και ήδη με το ψήφισμα που εγκρίθηκε την προηγούμενη εβδομάδα στο Στρασβούργο το πράξαμε αυτό. Ευχαριστούμε πολύ λοιπόν και ελπίζουμε να συνεχίσει να συνεχιστεί αυτή η συνεργασία μας. Colleagues, let's move on. Αγαπητοί συνάδελφοι, ας συνεχίσουμε, αλλά πρωτού συνεχίσουμε θα ακούσουμε τον κύριο Μιγκαρέλη, ο οποίος είναι ο διευθύνων σύμβουλος, μάλλον είναι ο διευθυντής, ο διευθυντής της Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης για τη Μέση Ανατολή και τη Νότια Γειτονία και σας υπενθυμίζω στις 5 και 4 θα πρέπει να ψηφίσουμε λόγω έλψης χρόνου αποφασίσαμε ότι η συζήτηση για την Κούβα θα πρέπει να αναβληθεί. Και προχωρούμε κατευθείαν στη συζήτησή μας με τον κύριο Μιγκαρέλη, από τον οποίο ζητώ να λάβει το λόγο για την Λιβύη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δύσκολο να περάσει κανείς από την Ουκρανία στη Λιβύη. Είναι πολύ διαφορετική η κατάσταση στις δύο χώρες. Θα προσπαθήσω όμως δύο μισή χρόνια μετά την δήλωση για την απελευθέρωση της Λιβύης που έγινε τον Οκτώβριο του 2011. Η Λιβύη παραμένει μια χώρα ασταθής όπου υπάρχουν εκδηλώσεις βίας κάθε είδους και όπου η πολιτική μετάβαση προχωράει με πολύ μεγάλα εμπόδια και δυσκολίες. Το πρόβλημα το οποίο βρίσκεται στην πηγή όλων αυτών των δυσκολιών είναι προφανώς η έλλειψη μιας πολιτικής ομαλοποίησης. Κυρίως γιατί δεν υπάρχει καμία συνένεση για ένα οδικό χάρτη σε σχέση με το πώς πρέπει να προχωρήσει αυτή η δημοκρατική μετάβαση. Επιμένω σε αυτό το σημείο γιατί είναι πάρα πολλοί παρατηρητές οι οποίοι εστιάζουν αποκλειστικά και μόνο στην κατάσταση ασφαλείας η οποία είναι φυσικά ανησυχητική. Πρέπει να κατανοήσουμε όμως ότι χωρίς μια επιτυχή πολιτική μετάβαση δεν υπάρχει παραμικρή δυνατότητα να λύσουμε οποιοδήποτε πρόβλημα ασφαλείας στη Λιβύη. Οι γεωγραφικές και εθνοτικές ομάδες στη Λιβύη έχουν αποδηθεί σε ένα αγώνα για τον έλεγχο των φυσικών πόρων και της εξουσίας και φυσικά αυτό ενισχύει την αστάθεια στη Λιβύη γιατί αυτές οι ένοπλες ομάδες ε, εξασφαλίσουν μια χαοτική κατάσταση, ενώ η κυβέρνηση είναι πάρα πολύ αδύναμη. Και ο Πρωθυπουργός ο κ. Ζιντάν δεν έχει δυνατότητα να επιβάλλει την τάξη και τον νόμο. Το Εθνικό Συμβούλιο είναι διηρημένο και πιο πολύ χρόνο δαπανά στον επιτίθεται κατά της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού του κ. Ζιντάν παρά να δίνει λύσεις. Υπάρχουν πολλοί ε, υπουργοί που ασκούν συνέχεια πιέσεις για οποιαδήποτε πολιτική απόφαση και η παρουσία των πολιτοφυλακών δημιουργεί απόλυτο χάος, υπάρχουν ε, απαγωγές, υποσπάθειε απαγωγών, δολοφονίες κτλ. Και κάθε φορά που πρόκειται να ληφθεί μια σημαντική πολιτική απόφαση από την κυβέρνηση, οι πολιτοφυλακές ασκούν με έμπρακτο τρόπο την πίεση αυτή και αυτό φυσικά επηρεάζει οποιαδήποτε απόφαση που μπορεί να ληφθεί από την κυβέρνηση. Αυτό έγινε με τον νόμο περί απομόνωσης. Ξέρετε ότι οι πολιτοφυλακές κατάφεραν να επιβάλλουν αυτή την νομοθεσία που εξασφαλίζει ότι όλοι οι πολιτικοί και οι υψηλοί αξιωματούχοι οι οποίοι στο παρελθόν ήταν τμήμα του καθεστώτος Καντάφη έχουν τον κίνδυνο να αποκλειστούν από οποιοδήποτε δημόσιο αξίωμα. Και από την άλλη πλευρά <clears throat> υπάρχει η σχεδόν απόλυτη απουσία κρατικού μηχανισμού. Πολλές χώρες έχουν ε, αδύνατες κυβερνήσεις και έλλειψη πραγματικού κράτους, αλλά στη Λιβύη δεν υπάρχει καν κρατικός μηχανισμός. Στα 42 χρόνια ε, διακυβέρνηση Καντάφη η δημόσια διοίκηση ήταν απόλυτα ανεμική. Δεν υπάρχει λοιπόν κρατικός μηχανισμός ο οποίος μπορεί να καλύψει την ανυπαρξία ή την αδυναμία της κυβέρνησης στη Λιβύη. Όλα αυτά έχουν σε αποτέλεσμα να είναι έφορες οι συνθήκες ώστε ο πληθυσμό να μην δίνει καμία εμπιστοσύνη στις πολιτικές αρχές και την εξουσία μέσα σε αυτό το θεσμικό και πολιτικό λοιπόν κενό κάθε είδους τυχοδιώκτες, κάθε είδους ένοπλες ομάδες και πολιτοφλέκες μπορούν να παίξουν ένα σημαντικό ρόλο. Ελλείψη λοιπόν ασφάλειας, βλέπουμε να υπάρχουν πολιτικές δολοφονίες και απαγωγές κυρίως στην περιοχή της ε, Βενγάζης. Γίνονται απαγωγές οι οποίες γίνονται για λίτρα αλλά και απαγωγές οι οποίες γίνονται για πολιτικούς λόγους. Υπάρχουν συνεχείς καταλήψεις ε, υπουργείων που δεν επιτρέπουν στα υπουργεία αυτά να λειτουργήσουν. Υπάρχουν επίσης καταλήψεις σταθμών φυσικού αερίου και πετρελαίου που κάνουν όλο και πιο δύσκολη και επισφαλή την οικονομική κατάσταση της χώρας αυτής. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν και σε αυτήν την κατάσταση τι μπορεί να κάνει η διεθνή κοινότητα και μέσα στη διεθνή κοινότητα τι μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Για να απλοποιήσω, έχω προσπαθήσει να εξηγήσω τι μπορούμε να προσπαθήσουμε τουλάχιστον να κάνουμε στον πολιτικό χώρο καταρχήν και μετά σε ό,τι αφορά τα θέματα ασφαλείας. Στον πολιτικό τομέα πρέπει προφανώς η συντακτική συνέλευση η οποία ε, εξελέγει πριν από μερικέ εβδομάδε να αρχίσει να εργάζεται. Αυτό δεν είναι εύκολο γιατί υπάρχουν πολλέ έδρε οι οποίε δεν καλύφθηκαν και έτσι αυτή η συντακτική συνέλευση είναι, ε, δεν είναι πλήρη και ορισμένοι θέλουν να εκμεταλλευτούν αυτή την κατάσταση για να ανατρέψουν την νομιμοποίησή τη. Δεύτερον, πρέπει να έχουμε ένα εθνικό διάλογο ο οποίος θα οδηγήσει σε μια εθνική συμφιλίωση πρέπει μέσα από τον εθνικό διάλογο οι κύριοι ηγέτες των, ε, κυρίως των κομμάτων και οι κύριοι ηγέτες της κοινωνίας των πολιτών να μπορέσουν να συζητήσουν με τα κύρια πολιτικά προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα η Λιβύη. Στη συνέχεια θα πρέπει να προσπαθήσουμε να πείσουμε τις αρχές, δηλαδή την κυβέρνηση και το εθνικό ε, συνέδριο να έχουν ένα περιεκτικό χαρακτήρα, δηλαδή να επιτρέψουν σε όλες τις πολιτικές δυνάμεις και όλες τις πτυχές της κοινωνίας των πολιτών να συμμετάσχουν στη διαδικασία εκπόνησης ενός, συστημα, ενός συντάγματος το οποίο μετά να τεθεί σε εφαρμογή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει καταλήξει σε κοινά μηνύματα, αυτό είναι πολύ θετικό. Έχουμε μπορέσει να συμφωνήσουμε για μερικά κοινά μηνύματα που θα στείλουμε στο σύνορο των πολιτικών δυνάμεων στην Λιβύη αλλά θα πρέπει να υποστηρίξουμε και με στεναρό τρόπο την αποστολή των Ηνωμένων Εθνών, την UNISMIL, η οποία κάνει ένα πολύ δύσκολο έργο, ένα άχαρο έργο σε δύσκολε συνθήκε και εκπροσώπω ε, των Ηνωμένων Εθνών, τα Ρεκμητρίφ, κάνει μια εξαιρετική εργασία και πρέπει να τύχει τη πλήρη υποστήριξή μα. Πρέπει επίση ω Ευρωπαϊκή Ένωση να έχουμε ένα συνεχή διάλογο με τον Πρωθυπουργό και τους κύριους Υπουργούς αλλά και το Εθνικό Συνέδριο για να μπορέσουμε να επηρεάσουμε τι επιλογές του. Θα πρέπει επίση να αντιμετωπίσουμε όλα τα προβλήματα που έχουν να κάνουν με τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα οποία δεν είναι εξασφαλισμένα, όπως ξέρετε, στη Λιβύη, ιδίω στις φυλακές, <clears throat> όπου υπάρχουν ακόμα κρατούμενοι πάρα πολλοί, πάρα πολλοί, οι οποίοι δεν έχουν δικαστεί ποτέ και είναι φυλαξισμένοι σε απαράδεκτε συνθήκε. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε και ένα διάλογο με τι αρχέ τη σε σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και επίση θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι έχουμε το μεγαλύτερο επίπεδο επαφών σε πολιτικό επίπεδο και επίπεδο υψηλών αξιωματούχων. Θα πρέπει να τεθεί το θέμα τακτικά στη Σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών και θα πρέπει να προχωρήσουμε στη διαπραγμάτευση της Συμφωνίας Πλαισίου που διακόπει στις αρχές του 2011 όταν έγινε η εξέγερση στη Λιβύη. Είναι απαραίτητο να συζητήσουμε και να διαπραγματευτούμε αυτή τη συμφωνία πλαίσιο για να ομαλοποιήσουμε τις σχέσεις μας με την Λιβύη, να θεωρηθεί μια φυσιολογική χώρα η Λιβύη και οι πολίτες της να μπορούν να έχουν μια συνολική άποψη του τι μπορεί να τους προσφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση και γι' αυτό το λόγο η διαπραγμάτευση αυτής της συμφωνίας πλαίσιου είναι το πιο σημαντικό εγχείρημα. Θέλουμε να επανέλθουμε στην Τράπεζα των Διαπραγματεύσεων το ταχύτερο δυνατό. Συνάντησα πριν από μερικές μέρες περίπου 30 Λίβιου της Βρυξέλλης για να τους εξηγήσω τι ακριβώς μπορεί να τους, πα, παράσχει η Ευρώπη μέσω αυτής της συμφωνίας και ότι είναι προς το συμφέρον τους να επανέλθουν στις διαπραγματεύσεις. Για τα θέματα ασφαλείας τι πρέπει να κάνουμε μαζί με τους κύριους διεθνεί εταίρους μας. Πρώτα απ' όλα να ε, αποστρατευτούν και να αφοπλιστούν οι πολιτοφυλακές. Αυτό είναι η πρώτη προτεραιότητα. Δεν είναι ιδιαίτερα εύκολο γιατί δεν έχουν ιδιαίτερο ε, ενδιαφέρον να αφοπλιστούν οι πολιτοφυλακές. Επίσης, μέσα με την διεθνή κοινότητα θα πρέπει να ασχοληθούμε με την κατάρτιση της ε, αστυνομίας και τη δημιουργία ενός εθνικού στρατού. Υπάρχουν πολλές χώρες οι οποίες μέσα στο σύμφωνο των G8 μαζί με τον ΝΑΤΟ εργάζονται για την καλύτερη κατάρτιση των στρατιωτικών. Στην ε, Φιλιβή πρέπει να, να εκπαιδευτούν 15.000 στρατιώτες από την Ιταλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία, τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Τουρκία. Ελπίζουμε λοιπόν ότι θα καταστεί δυνατό μέσα στους επόμενους μήνες να εκπαιδευτεί και να εξοπλιστεί ο στρατός αυτός για να υπάρχει τουλάχιστον ένα ένας εμβριώδης <clears throat> στρατό στη Λιβύη που μπορεί να εξασφαλίσει την ειρήνη. Προσπαθούμε επίσης να εξασφαλίσουμε και την ε, εκπαίδευση της αστυνομία, αλλά είναι δύσκολο να βρούμε σταθερούς και αξιόπιστους ε, συνομιλητές στην πλευρά της Λιβύης. Μετά πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι θα έχουν τη βοήθειά μας για να ελέγχουν τα σύνορά τους. Υπάρχει η αποστολή EUBAM και υπάρχουν περίπου 50 Ευρωπαίοι εμπειρογνώμονες οι οποίοι βοηθούν τις αρχές της Λιβύης να ε, εκπαιδεύσουν τους φύλακες στο σύνορο. Θα είναι δύσκολο, δεν μπορούμε 50 εμπειρογνώμες να το πετύχουμε. Οι Λίβοι έχουν 6.000 ε, ε, μίλια σύνορα, 4.000 επίγεια και 2.000 θαλάσσια και πρέπει να συνεργαστούμε και με τους Αμερικανούς. Πέρα από τον έλεγχο των σύνορων θα πρέπει να τους βοηθήσουμε να ελέγξουν καλύτερα τις αποθήκες όπλων. Ξέρετε ότι υπάρχουν πολύ σημαντικές ε, ποσότητες πυρομαχικών και όπλων στη Λιβύη. Θέλουμε να τους βοηθήσουμε να ελέγξουν αυτά τα όπλα και να ενισχύσουμε την ασφάλεια στη Λιβύη και να αποφύγουμε έτσι ώστε η παρουσία η μαζική αυτών των όπλων αποστεθροποιήσει το σύνολο του Μαγκρέμ και του Σαχέλ όπως το είδαμε στο Μαλί πριν λίγους μήνες. Ε, προσπαθούμε και οι Βρετανοί επίσης και οι Αμερικανοί παίζουμε και εμείς στα πλαίσια των δυνατοτήτων των ρόλων μας. Δεν θα μακρηγορήσω πρόεδρε. Πρέπει να συνεργαστούμε με τους γείτονες της χώρας αυτής. Συνεργαζόμαστε λοιπόν σε περιφερειακό επίπεδο με τους Λίβιους, με όλες τις γειτονικές χώρες, το Μαλί, τη Μαυριτανία, το Τσάδ, το Νίγηρα και θα θέλαμε επίσης και οι χώρες του Μαγκρέμπ, η Αλγερία, το Μαρόκο και η Τινησία να εμπλακούν και αυτοί. Δεύτερον θα πρέπει να ενισχύσουμε την συνεργασία και το συντονισμό των διεθνών εταίρων. Αυτό θα είναι ο στόχος της συνάντησης που θα διεξαχθεί την Πέμπτη στη Ρώμη σε υπουργικό επίπεδο. Ελπίζουμε αυτή η υπουργική συνάντηση στη Ρώμη να επιτρέψει να ξεκινήσει επιτέλους η πολιτική μετάβαση με την στήριξη της διεθνούς κοινότητας. Ελπίζουμε επίσης ότι η συνεδρίαση αυτή στη Ρώμη θα μας επιτρέψει να κατανείμουμε καλύτερα τις αρμοδιότητες στα πλαίσια της διεθνούς κοινότητας σε σχέση με αυτά τα οποία κατά προτεραιότητα μένει να γίνουν για να δώσουμε εγγυήσει για τη σταθερότητα και την ασφάλεια σε αυτή τη δυστυχή χώρα. Ευχαριστώ. Ο Σερ Ρόμπερτ. Χαίρομαι να σας βλέπω να προεδρεύετε. Ε, ήταν πολύ σημαντική η επιλογή των ε, ε, κοσμητόρων, λέει ο κύριος Άτκιν. Σε πάση περιπτώσει, τρεις ερωτήσεις έχω να θέσω. Βλέποντας ότι το κοινοβούλιο δεν λειτουργεί όπως θα θέλαμε, βλέπετε εσείς να υπάρχει μια κάποια επιθυμία για αυτό το οποίο ονομάζουμε ισχυρή διοίκηση κεντρική, ένας άλλος δικτάτορας δηλαδή σε εισαγωγικά που θα, φέρει, ε, θα ενώσει τη χώρα. Το πιστεύουν κάποιοι αυτό. Δεύτερον, είπαμε ότι η κοινοβουλευτική διαδικασία δεν λειτουργεί σωστά. Τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να καθοδηγήσει αυτές τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες, τι know-how δίδουμε στους Λιβύους για να το πετύχουν αυτή τη φορά. Και μια τελευταία ερώτηση θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι δεν είναι τόσο σημαντική σε σχέση με την απώλεια της ζωής των δικαστών και την ανεξαρτησία των δικαστών κτλ. Στη Λιβύη υπάρχουν τεράστιοι αρχαιολογικοί ε, χώροι, πάρα πολύ σημαντικοί στην Κυριναϊκή, Υπάρχουν επίσης και στρατιωτικά νεκροταφεία από τους παγκόσμιους πολέμους. Όλα αυτά έχουν μεγάλη σημασία με τον ένα τρόπο ή τον άλλο. Γίνεται κάτι για την προστασία αυτών των ιστορική σημασίας χώρων. Ευχαριστώ Μίλαν Μόν. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Δεν άκουσα την αρχή της παρουσίασής σας παρά μόνο στο τέλος. Αν κατάλαβα καλά, πιστεύετε ότι η συνεδρίαση της Ρώμης θα βοηθήσει έτσι να συντονιστούν καλύτερα οι βασικοί εταίροι της διεθνούς κοινότητας που συνεργάζονται στη Λιβύη. Ποιο είναι το επίπεδο συνεργασίας των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συνεργάζονται γιατί εδώ άκουσα έναν συνάδελφο να μιλά, να διαμαρτύρεται για την έλλειψη συνεργασίας από πλευράς κάποιων κρατών μελών και για μια γενικότερη έλλειψη συνεργασίας. Θα ήθελα να μας αναλύσετε λίγο αυτό το θέμα. Πάρα πολλοί συμφωνούν ότι το θέμα της Λιβύης στην ουσία οδηγεί σε μια τεράστια βαλκανοποίηση της χώρας είναι μια χώρα η οποία αποτελείται από φιλετικές ομάδες οι οποίες έχουν διαιρεθεί μεταξύ τους και οι οποίες δυσκολεύονται να ακολουθήσουν μια θεσμική μορφή συνεργασίας. Και ο Καντάφη κατάφερε με, την σιδερένια του γροθιά να τα αυτά τα συστήματα, αλλά τώρα πλέον είναι πάρα πολύ δύσκολο να διασφαλιστεί η ενότητα του παρελθόντος. Ίσως αυτή είναι μια παρατήρηση πάνω στην οποία να κάνετε κάποια σχόλια. Αν πράγματι είναι αδύνατο τελικά να καταλήξει η χώρα αυτή σε ένα αίσθημα ενότητας ανάμεσα σε φυλές οι οποίες όχι μόνο μεταξύ τους δεν συνεννοούνται αλλά και στο εσωτερικό τους υποφέρουν από οικογενειακού τύπου διαιρέσεις. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε. Πρόεδρε, και εγώ να ευχαριστήσω τον κύριο Μιγκαρέλη να τον ρωτήσω πιο πολλές λεπτομέρειες σε ό,τι αφορά το κοινοβούλιο που θα πρέπει να στρωθεί στη δουλειά. Μου φαίνεται ότι η δυσκολία δεν έγινε τόσο πολύ στον ότι το κοινοβούλιο δεν θέλει να δουλέψει, αλλά ότι δεν μπορεί να δουλέψει. Λιθοβολήθηκε, αναγκάστηκε να μετακομίσει σε ένα ξενοδοχείο. Ο πρόεδρος του κοινοβουλίου, κ. Σαχμέν, δέχεται διαρκώς επιθέσεις και αναρωτιέμαι τι μπορεί παραπάνω να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να συνδράμει και να βοηθήσει το Κοινοβούλιο της Λιβύης να αντιμετωπίσει την κατάσταση και να ρωτήσω και το θέμα των πόρων. Υπήρχε γενικώ η ελπίδα πριν από ένα-δύο χρόνια ότι τα έσοδα από το πετρέλαιο και από το αέριο θα μπορούσαν να χρηματοδοτήσουν την ανοικοδόμηση της χώρας. Και αυτό δεν φαίνεται να συμβαίνει, δεν φαίνεται. Φαίνεται ότι υπάρχει μάλλον μεγάλη σύγκρουση. Τι πόρους λοιπόν έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση και πώς οι πόροι αυτοί συγκρίνονται σε σχέση με τους πόρους που υπήρχαν κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης. Γιατί λοιπόν δεσμευόμαστε λιγότερο υπέρ της Λιβύης Γιατί ενώ μπορέσαμε, ότι θα μπορέσουμε να κερδίσουμε τον πόλεμο, δεν μπορούμε να κερδίσουμε και την ειρήνη. Ο Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για τις ε, παρουσιάσεις σας πάρα πολύ ενδιαφέρουσες. Θα ήθελα να επανέλθω σε αυτά που είπε ο συνάδελφος ε, Μίλαν Μόν σε ό,τι αφορά τις ε, ομάδες οι οποίες προσπαθούν να διασφαλίσουν ό,τι περνάει από το χέρι τους. Ισχύει αυτό. Και κατά δεύτερον, έχω την εντύπωση ότι η διεθνής κοινότητα όλο και πιο πολύ εγκαταλείπει πράγματα. Είτε για την Ουκρανία μιλάμε, είτε για τη Συρία. Για την καταστροφή των χημικών όπλων. Αλλά έχω την εντύπωση ότι η Λιβύη έχει εξαιρεθεί από τον χάρτη των χωρών με κρίση και ότι πολύ απλά την έχουμε αφήσει εκτός. Ισχύει αυτό. Uh, Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Μιγκαρέλη. Ευχαριστώ να απαντήσω πρώτα στον Sir Robert. Αν υπάρχει θέληση για μια ισχυρή η ηγεσία στη Λιβύη. Ναι, υπάρχει σαφή θέληση σήμερα στη, στη Λιβύη για κάτι τέτοιο, γιατί όπως μπορείτε να φανταστείτε, ο πληθυσμός έχει πια βαρεθεί να ζει σε μια τόσο χαοτική κατάσταση. Οι συνθήκες διαβίωσης έχουν επιδεινωθεί λόγω αυτού του χάους και είναι φανερό ότι υπάρχει μεγάλη θέληση για να υπάρξει επιστροφή στον νόμο και την τάξη. Μπορούμε να έχουμε νόμο και τάξη χωρίς μια δικατορία. Το ελπίζω. Πιστεύω. Νομίζω ότι οι εμπειρίες μετάβασης σε πολλές χώρες του κόσμου δείχνουν ότι ακόμα και στις χειρότερες συνθήκες και η Λιβύη είναι πραγματικά στις πιο δύσκολες των δύσκολων καταστάσεων γιατί δεν υπάρχει μονάχα η έλλειψη μιας πολιτικής τάξης υπάρχει απόλυτη απουσία κρατικού μηχανισμού. Αν συνδυάσετε τα δύο βλέπετε ότι είναι πραγματικά οι χειρότερε των χειροτέρων συνθήκων για να υπάρξει μια διαδικασία μετάβαση στη δημοκρατία. Παρ' όλα αυτά αυτοί που κάναν την επανάσταση στη Λιβύη σίγουρα θέλουν να επιτύχουν νόμο και τάξη στη Λιβύη χωρί όμω να εγκαταστήσουν ένα νέο δικτάτορα. Θα χρειαστεί χρόνο αυτό λοιπόν, αλλά θα το πετύχουμε. Το δεύτερο ερώτημα. Πώς θα τους ε, καθοδηγήσουμε και θα τους βοηθήσουμε. Και εδώ έρχομαι στο ερώτημα του κυρίου Βάτσον. Έχουμε δώσει μετά από το τέλος της σύγκρουσης στη Λιβύη 130 εκατομμύρια ευρώ σε τομείς όπως η δημιουργία δημόσιου, δημόσιας διοίκησης, βελτίωση της κατάστασης αστυνομίας, μεταρρύθμιση του δικαστικού σώματος, ενίσχυση της ανάπτυξης της κοινωνίας των πολιτών. Αλλά φυσικά δεν είναι εύκολο να εφαρμόσουμε όλα αυτά τα σχέδια, γιατί όπως σας είπα δεν έχουμε ενώπιον μας σταθερούς και αξιόπιστους συνομιλητές. Δεν υπάρχει μια δημόσια διοίκηση όπως υπήρχε πριν από 30 χρόνια στην Τσεχοσλοβακία ή στην Πολωνία ή πριν από 15 χρόνια στα Δυτικά Βαλκάνια. Δεν υπάρχει τίποτα σε επίπεδο δημόσιας διοίκησης, γι' αυτό είναι πολύ δύσκολο για τους εμπειρογνώμονές μας να κάνουν τα σχέδια υποστήριξης τους αλλά προσπαθούμε να προχωρήσουμε όσο μπορούμε περισσότερο με αυτά τα σχέδια για να τους καθοδηγήσουμε στο δρόμο της μετάβασης. Υπάρχει και μια ανάγκη να προστατεύσουμε τις μειονότητες και αυτό μας απασχολεί και ο στόχος μας είναι να εξασφαλίσουμε ότι όλοι αυτοί οι οποίοι είναι κρατούμενοι χωρίς να έχουν τύχη δίκαιας δίκης θα μπορέσουν είτε να δικαστούν πράγματι ή να απελευθερωθούν το ταχύτερο δυνατό. Για τον κύριο Μιλανμόν αν υπάρχει πρόβλημα συντονισμού με τα κράτη-μέλη στη Λιβύη. Για να είμαι απόλυτα ε, ειλικρινής θα πρέπει να αγωνιστούμε για να μπορέσουμε να πετύχουμε κάποιο βαθμό ε, συντονισμού και για να είμαι πάλι ειλικρινής δεν είναι καθόλου παράξενο κάτι τέτοιο. Υπάρχει φυσικό αέριο και πετρέλαιο, υπάρχουν αυτοί οι οποίοι ενδιαφέρονται για μεγάλα συμβόλαια στον τομέα αυτό και επομένως υπάρχουν πολλές ε, διαμάχες για τα θέματα αυτά. Πρέπει να σεβαστούμε λοιπόν τον ανταγωνισμό για αυτά τα συμβόλαια, αλλά συγχρόνως να εξασφαλίσουμε ότι τα κράτη-μέλη και τα ευρωπαϊκά όργανα θα μπορέσουν να έχουν καλύτερο συντονισμό για να προσπαθήσουμε να έχουμε μεγαλύτερη επιρροή στην πολιτική μεταρρύθμιση, αλλά και να εξασφαλίσουμε την ασφάλεια. Έχουμε κάνει κάποια πρόοδο δεν έχουμε μια κατάσταση που είναι απόλυτα ικανοποιητική. Θα πρέπει να συνεχίσουμε τον αγώνα μας και πιστεύω ότι με καλή θέληση και ενεργητικότητα μπορούμε να καταλήξουμε σε μια βελτίωση της κατάστασης. Έχετε δίκιο όταν λέτε ότι η διαίρεση σε φυλέ και φάρες είναι πολύ σημαντική. Γιατί ο Καντάφη κατάφερε να ενώσει όλες αυτές τις φυλέ. Γιατί είναι πιο εύκολο για ένα δικτάτορα να κάνει τις φυλές να συμφωνήσουν από ότι να λειτουργήσει ένα δημοκρατικό καθεστώς. Αυτό δεν εκπλήττει κανένα. Έχετε λοιπόν πολλές φυλές οι οποίες μάχονται εναντίον η μια της άλλης, φυλές που είναι οργανωμένες σε γεωγραφικό επίπεδο. οι, οι πολιτοφυλακές της Ίνταν και της Μιντάσα είναι πάρα πολύ σημαντικές. Ξέρετε ότι υπάρχουν οι αμαζίγοι του Αρέκ, Ντεμπού, οι οποίοι δεν θελήσαν να συμμετάσχουν στο δημοψήφισμα για το Σύνταγμα μάλλον το δημοψήφισμα για τη συντακτική συνέλευση. Υπάρχουν λοιπόν πολλές δυσκολίες με τις διάφορες φυλές στη Λιβύη. Αυτό κάνει όμως το σούτον μάλλον σημαντικό, το να υπάρξει μια περιεκτική διαδικασία και όλα αυτά μας δείχνουν πόσο η κυβέρνηση και το κοινοβούλιο, αν θέλουν κάτι συγκεκριμένο να πετύχουν, θα πρέπει να προσπαθήσουν να είναι περιεκτικοί και να εξασφαλίσουν ότι όλοι συμμετέχουν στην δημοκρατική διαδικασία. Είπε ο κύριος Βουατσόν ότι το Κοινοβούλιο είναι κάτω από συνεχή επίθεση. Υπάρχει πράγματι απειλή των πολιτοφυλακών εναντίον του Κοινοβουλίου που είναι το Εθνικό Συνέδριο και της κυβέρνησης αλλά και μέσα στο Κοινοβούλιο πολεμούν οι μεν τους δε συνέχεια και ακόμα και σε καθημερινή ε, βάση εκτοξεύουν απειλές κατά του Πρωθυπουργού. Πρέπει να στήσουμε λοιπόν του κοινοβουλευτικού να είναι πιο υπεύθυνοι και να δρούν προ το συμφέρον του λιβικού λαού. Ο κ. Καραστόφλερ. Μπορεί η Λιβύη να θεωρηθεί ακόμα προτεραιότητα της ε, Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι. Γιατί αν γίνει μια μαύρη τρύπα αύριο, αυτό θα έχει άμεσες συνέπειες για την Ευρώπη σε ό,τι αφορά πρόσφυγες, παράνομη μετανάστευση οργανωμένο έγκλημα. Δεν έχουμε λοιπόν καμία επιλογή παρά να κρατήσουμε την Λιβύη ψηλά στην ημερήσια διάταξή μας και αυτό κάνουν οι πολιτικοί μας ηγέτες. Ευχαριστώ. Να συμπληρώσω κάτι εδώ για τις αρχαιότητες και την αρχαιολογική κληρονομιά. Κοιτάξτε, δεν μιλάμε, δεν συζητάμε το θέμα αυτό. Δεν σας λέω ότι το θέμα δεν είναι σημαντικό. Πρέπει να στρέψουμε την προσοχή μας και σε αυτό. Θυμάμαι ότι εδώ και δύο χρόνια όταν συζητούσαμε τη συμφωνία πλαίσιο με το τέος καθεστώς είχε τεθεί το θέμα ε, των πολιτιστικών των χώρων κτλ. Και η αντιπολίτευση μας είχε βοηθήσει να διαχειριστούμε τους χώρους αυτούς. Σήμερα όμως είναι ένα θέμα το οποίο με κάθε ειλικρίνεια δεν τίθεται όταν συζητάμε με τους Λιβύους. Συμφωνώ μαζί σας όμως ότι είναι κάτι το οποίο πρέπει να μας απασχολήσει. Ευχαριστώ. Ελπίζω να ελεγχθεί η κατάσταση εκεί γιατί σε άλλα μέρη δεν ελέγχεται σας εύχομαι ό,τι καλύτερο και εύχομαι να τα ξαναπούμε σύντομα. So, uh, dear friends, we have votes. Λοιπόν, έχουμε ψηφοφορίες σε 10 λεπτά. 5 και 4 και κάνουμε διάλειμμα μέχρι τις 5 και 4. Damen und Herren, αγαπητοί συνάδελφοι, επιτρέψτε μου να περάσω στο σημείο 7 της ημερήσιας διάταξης ψηφοφορία για την έκθεση προόδου για την Τουρκία. Η συγγήτρια είναι η κυρία Κυρία Ομινρόιτεν, έχετε κάποια σχόλια να κάνετε. Πρόεδρε, ελπίζω οι σοσιαλιστές να τηρήσουν τις συμφωνίες που κάναμε για αρκετά κρίσιμα σημεία. Και ελπίζω λοιπόν να τηρήσουν τις συμφωνίες αυτές. Γιατί μέσα σε μία ώρα σήμερα το μεσημέρι έχει αλλάξει λίγο ε, η τάση που επικρατεί. Εδώ σε αυτό το κοινοβούλιο πρέπει να υπάρχει δούνε και λαβίν. Δούνε και λαβίν. Τι σημαίνει αυτό να κάνουμε και συμφωνίες. Και οι συμφωνίες θα πρέπει να τηρούνται, θεωρώ. Πρόεδρε, είναι η πρώτη φορά που μου συμβαίνει αυτό το πράγμα. Και ελπίζω... Ελπίζω να μην ε, υποκύψουν τελικά στα βήματα αυτά, τέλος πάντων, που είναι απαράδεκτα. Ως σοσιαλιστές είχαμε κάνει μια συνεδρία ομάδα εργασία πριν από τη συνεδρίασή μας και δημοκρατικά καταλήξαμε σε μια διαφορετική απόφαση από αυτή που είχε γίνει στη συνάντηση των σκι... σκιωδών συγητών. Γι' αυτό υπάρχει μια διαφορετική θέση από τη θέση που είχε συμφωνηθεί αρχικά, αλλά νομίζω ότι κάτι παρόμοιο είναι και σε άλλες ομάδες. Ευχαριστώ. Είναι ένας χώρος ελευθερίας, ακόμα και αν αυτό δεν βολεύει πάντα, λέει ο πρόεδρος και ο καθένας μπορεί να πράξει ελεύθερα αυτό το οποίο θέλει. Ψηφοφορία. Τροπολογία 41. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 43. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 47 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 52 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβασκή 2 υπέρ κατά αποχές δεκτή Τροπολογία 57. Με την κατάλληλη τροποποίηση υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 59 και 60 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 61 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 63 62 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 63 έχει αποσυρθεί συμβαστική 3 υπέρ κατά αποχές δεκτή 77 υπέρ υπέρ είπα κατά αποχέ απορρίπτεται. 80 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 82 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 86 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 4 υπέρ κατά αποχές δεκτή 87 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 92 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 100 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 103 υπέρ με προφορική τροποποίηση υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 105 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 100 107 λέει ο πρόεδρος. 104 καλύτερα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 106 υπέρ κατά αποχές. Νομίζω ότι εγκρίνεται, αλλά ας ελέγξουμε. 106. Εγκρίνεται. Συμβαστική 6 υπέρ. Είχαμε την 107 προηγουμένως. Α, 107 μάλιστα υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 6 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 7 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 126 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 131 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστή 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 132 υπέρ κατά αποχές απολύτω. Όχι, όχι. 135 υπέρ κατά αποχές. Νομίζω ότι την δείτε να ελέγξουμε. Να ich, meine ich, meine Ja, απορρίφθηκε, απορρίφθηκε. Ja, dann hat Έλεξη ψηφοφορία. Α, κάτι λάθος μετρήσαμε, λέει ο Πρόεδρος. Απορρίπτεται με σαφή διαφορά. Και περνάμε λοιπόν στην 136, υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Και τώρα λοιπόν... 141. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 144. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 160 υπέρ. 160 υπέρ. Για την 144. Αφού ψήφισαν όχι οι σοσιαλιστές. Έλεγχος. Έλεγχος για την 144. Ναι, Look, but we cannot use the check for changing the Ναι, κοιτάξτε, αλλά δεν μπορούμε να χρησιμοποιούμε τον έλεγχο για να αλλάξουμε θέση οποιοδήποτε. Δεν είναι αποδεκτό αυτό το κόλπο. Είναι καλό το κόλπο, δεν λέω. Να το θυμηθώ και την άλλη φορά. Πέρας ψηφοφορίας. Αλλά δεν βοήθησε. Και πάλι. Και περνάμε στην 160. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 145 υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 9 υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. 146 υπέρ. Κατά. Άποχες απορρίπτεται. Και τώρα περνάμε λοιπόν. 150 υπέρ. Κατά. Άποχες. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 158 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 162. υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 10 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 170 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Α, όχι. Να ελέγξουμε παρακαλώ την 170. Δεν ήμουν συγκεντρωμένος, το ομολογώ. Η ηλεκτρονική, ηλεκτρονικός έλεγχος. Δεν το πρόσεξα. Πέρα ψηφοφορίας. 8 υπέρ, 36 κατά. 173 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 174. 173 εγκρίθηκε. Ζητείτε έλεγχος. Now we Για να δούμε τη δύναμη των φιλεύθερων, λέει ο Πρόεδρος.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 Ναι, είναι ένα πρόβλημα αυτό με την κατανόηση μεταξύ Γερμανών και Ελλήνων. «179 υπέρ». Κατά. Άποχες. Απορρίπτεται. Συμβαστική 11 υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. 179. υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Απορρίπτεται. Απορρίπτεται διορθώνει ο Πρόεδρος. Απορρίφθηκε. Και περνάμε τώρα στη συμβαστική 12, υπέρ. Μα μόλις ψηφίσαμε, λέει ο πρόεδρος. Ναι, ξεχάσαμε την 189. Την 191. Απορρίφθηκε η 189, η 191 υπέρ. Κατά. Αποχές δεν βοήθησε. Δεν βοήθησε. Συμβαστική 12 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 196 υπέρ. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 199 υπέρ. Κατά. Άποχες απορρίπτεται. Η 200 υπέρ. Κατά. Άποχες. Απορρίπτεται. Η 201 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η 202 υπέρ. Κατά. Άποχες. Απορρίπτεται. Συμβαστική 13 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 210 υπέρ. Κατά. Αποχές. Να το ελέγξουμε παρακαλώ. Δεν είναι σαφές το αποτέλεσμα. Για τη 210. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται 20 ψήφοι υπέρ, 26 ψήφοι κατά. 211 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 212 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 14 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η 232 υπέρ. 223 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 224 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 225 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 226 υπέρ. Κατά άποχες απορρίπτεται. 234 υπέρ. Κατά άποχες απορρίπτεται. Συμβαστική 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 230 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 231-232 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Και εδώ είχαμε έναν ε, συγγραφέα που πήρε διπλά έσοδα συγγραφής. 233 υπέρ. Α, έχει καταπέσει. Και αυτή καταπίπτει, μάλιστα. Mein Päckchen ist die andere äh, Seite herum Έχω αλλάξει σελίδα στο πακετάκι μου εδώ. Ε, Κάποιο έχει βάλει ένα από τι σελίδε μου. 238 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 239 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 240. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Εγκρίνεται. 242 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 243 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 246 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 16 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 250 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 16α υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 261 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 266 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 267 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 276 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 275 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Απορρίπτεται, απορρίπτεται, απορρίπτεται, διορθώνει ο πρόεδρος. Η 275 Την 269 την έχουμε ψηφίσει ακόμα. 268. Υπέρ. 268 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 269 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 270 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 271 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 272 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 273 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 274 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 277 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 278 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 279 υπέρ. Κατά αποχές, απορρίπτεται. 280-281 υπέρ. Κατά. Άποχες. Απορρίπτεται. 282 υπέρ. Κατά. Άποχες. Απορρίπτεται. 283 υπέρ. Κατά. Άποχες. Απορρίπτεται. 284 υπέρ. Κατά. Άποχες. Απορρίπτεται. 285 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 286 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 287 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 288 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 289 υπέρ. Κατά. Για την 289. Έλεγχος παρακαλώ. 13 υπέρ, 33 κατά απορρίπτεται. 292 υπέρ. Α, 290. 290 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 292 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 294 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 295 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 296 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται 297 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται 298 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται 299 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Η 300 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται 301 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται 302 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται 303 υπέρ. Κατά. Άποχες. Απορρίπτεται. Η 305 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 306 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 307 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η 309 υπέρ. Κατά. Άποχες. Έλεγχος παρακαλώ. Για την 309. Έλεγχος. Πέρας ψηφοφορίας. 11 υπέρ, 37 κατά, απορρίπτεται. 310 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 311 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρι... ε, απορρίπτεται. Έλεγχος για την 311. Για την 311 απορρίφθηκε. Α, άλλαξαν στάση οι σοσιαλιστές, αλλά μόνο εν μέρη, λέει ο πρόεδρος. Πέρα ψηφορίας. 11 υπέρ, 32 κατά. Η 312 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 314 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 315 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 316 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 17 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 326. Μποσκούρτ. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 327 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 18 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 337 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Το κύριο Σταφ. Ναι, πρόεδρε για την 338. Θα ήθελα να ζητήσω να υπάρξει μια καταδιέρεση ψήφος. Καλούμε, λέμε, το επόμενο Κοινοβούλιο και την επόμενη Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διασφαλίσουν την συνέχεια της δυνατότητας πρόσβασης, ένταξης μάλλον, της διαδικασίας μάλλον την οποία ε, ε, ακολουθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Τουρκία εδώ και αρκετά χρόνια. Και μετά το υπόλοιπο κομμάτι. Κοιτάξτε, έχουμε συγκεκριμένους κανόνες εδώ αν θέλει κάποιος να ζητήσει μία καταδιέρεση ψήφο πρέπει να το ζητήσει νωρίτερα. Ο κύριος Νταφ ξέρει ότι είμαστε κατά της τροπολογίας. Αν θέλει να ιτηθεί δύο φορές ας δεχθούμε το αίτημά του. Äh, äh, er. Andrew, I'm Καταλαβαίνω την απόψή σου, αλλά πρέπει να σεβαστώ τους κανόνες. Αν απορρίφθηκε λοιπόν, απορρίφθηκε το αίτημα αυτό. Ας ψηφίσουμε λοιπόν ποιος είναι υπέρ του 338. Κατά. who accepts who is in Υπέρ, υπέρ λέει ο Πρόεδρος. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η τροπολογία 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 5. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 6. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος παρακαλώ. Για την έξη. Πέρας ψηφορίας. 13 υπέρ, 34 κατά. Απορρίπτεται. 7 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 8 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 9. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 10. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 11. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 12. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 13. 13. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 14. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος παρακαλώ. Για την 14. Πέρα geschlossen. Πέρα 12 υπέρ, 34 κατά. Πάντα είναι πολύ λανθασμένη η εκτίμησή μας σήμερα. Η 16 υπέρ. Α, η 15 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 16 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 17 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 18 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 19 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 20 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 21. Έλεγχος για την 20. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 20. Πέρας ψηφοφορίας. 35 ψήφοι υπέρ, 13 κατά, εγκρίνεται. 23 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 24-25 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 26 υπέρ, κατά, αποχές, θα έλεγα ότι εγκρίνεται εκτός ε, και αν συμμετείχε το ΕΛΚ. Έναρξη ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. Πέρας ψηφοφορίας. 19 ψηφί, 30 κατά. 26. 26. Α, μάλιστα. 27. Υπέρ. Κατά απόχέ απορρίπτεται. 28. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται.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 Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται η έκθεση με 36 ψήφους υπέρ, 8 κατά, 5 αποχές. Σας ε, συγχαίρω κυρία Συγκητρία. Äh, Ευχαριστήσω, Ρία, γιατί το, την έκθεση αυτή την, ε, το, το παρακολουθήσατε εδώ και καιρό και πάντα συγκεντρώνεις μεγάλες πλειοψηφίες σε αυτό το πάρα πολύ δύσκολο θέμα και Θα ήθελα να σε ευχαριστήσω για όλα αυτά τα χρόνια που έχεις αναλάβει αυτό το έργο, γιατί θα είναι και η τελευταία έκθεση που αναλαμβάνει για την Τουρκία. Κοιτάξτε, Πρόεδρε, ποτέ δεν ήταν βαρετή αυτή η στιγμή, αυτή η εργασία του να είναι κανεί εισηγητής για την Τουρκία. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όμω και του συναδέλφου μου. Όχι μόνο για σήμερα, αλλά ιδιαίτερα σήμερα, που επιτέλους ακολουθήσαμε αυτά επί των οποίων συμφωνήσαμε τις τελευταίες εβδομάδες. Ήταν λοιπόν κρίσιμη σημασία. Όλα αυτά τα χρόνια που έκαναν την έκθεση πρόοδου για την Τουρκία να καταφέρουμε να βρούμε μια συμφωνία στο Κοινοβούλιο. Μια ειλικρινή συμφωνία που θεωρεί την Τουρκία υποψήφια, αλλά διαπραγματευόμαστε μαζί της και την αντιμετωπίζουμε με ανοιχτό και δίκαιο τρόπο. Υπάρχουν πολλά σημεία κριτικής, ιδιαίτερος φέτος, αλλά πάντα με ανοιχτό και δίκαιο τρόπο και ελπίζω να υπάρξει μεταρρύθμιση της χώρας, γιατί αν θέλουν ευημερία χρειάζονται κατεπηγόντως μεταρρυθμίσεις. Να ευχαριστήσω εκ νέου όλους τους συναδέλφους, ιδιαίτερα στη Μαρία και όλους τους υπόλοιπους, που σε κάποια δύσκολα ζητήματα καταφέραμε να συνεννοηθούμε. Σας ευχαριστώ. Δεν χρειάζεται να μας ευχαριστήσεις, ε, γιατί πολλοί από εμά απλώς φοβόμασταν να ψηφίσουμε διαφορετικά από σένα. Το επόμενο σημείο της της διάταξης. Για τις ε, εκπομπές ως τμήμα της ευρωπαϊκής διπλωματίας. Ε, θέλω να δώσω το λόγο στον αθλητικό εισηγητή, τον κύριο Γκράμζο Βότσον. Ε, Συγγνώμη δεν μπόρεσα να με παρών την προηγούμενη εβδομάδα στη συνεδρία της Επιτροπής λόγω ενός ατυχήματος το οποίο με έβαλε στο νοσοκομείο αλλά το ποδήλατό μου δεν έπαθε τίποτα. Θα χαρούν να το ακούσουν αυτό οι συναδελφοί μου. Θέλω ευχαριστώ τον κύριο Φαν Μπάλεν και τους χειόδης συζητητές. Υπάρχουν μερικές τροπολογίες συμβασμού. Όλες υποστηρίζονται από μένα. Πέντε προφορικές τροποποιήσεις επίσης και δεν έχω καμία αντίρρηση στις δύο έως πέντε. Υπάρχει ένα πρόβλημα για τον τίτλο αυτής της έκθεσης και από ό,τι κατανοώ, από τη στιγμή που έχει προταθεί από το Προεδρείο μιας Επιτροπής ο τίτλος και έχει γίνει δεκτός από την Συνέλευση των Προέδρων, δεν μπορεί να τροποποιηθεί με τροπολογία. Αλλά μπορεί να αλλάξει μόνο από τη Συνέλευση των Προέδρων. Θα ήθελα να σα ζητήσω λοιπόν να ζητήσετε από τη Συνέλευση των Προέδρων να ζητήσετε να αλλάξει ο τίτλο σε ένα νέο τίτλο ο οποίο έχει συνέλευση Οπότε θα είναι σχέδιο συστάσεως στο Συμβούλιο των Κομισιών και την Υπηρεσία Εξωτερικών Δράσεων για το ρόλο των μέσων ενημέρωσης σε ό,τι αφορά την προβολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των αξιών της. Εάν θέλετε λοιπόν να εγκρίνει η Επιτροπή μας μια τέτοια αλλαγή και να τη συνιστήσει προς τη συνέλευση των Πρόεδρων, θα μπορέσουμε να βρούμε έτσι μια συμβαστική λύση για όλους. Σας ευχαριστώ, θα το προσπαθήσουμε λέει ο Πρόεδρο. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος λόγος να μην ε, προχωρήσουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Είναι απλώς μια προφορική, μια λεκτική κατά κάποιο τρόπο παρεξήγηση η οποία μπορεί να δημιουργηθεί από τον τίτλο αυτόν. Και θα δώσει και δουλειά σε κάποιους. Ποιος υποστηρίζει τον νέο αυτό τίτλο που ανέφερε ο συγητής, παρακαλώ σηκώστε το χέρι σας κατά αποχές έχει γίνει δεκτός ο νέος τίτλος. Και περνάμε στην συμβιβαστική 4. Ψήφι υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 58 και 59 υπέρ. Κατά αποχές έλεγχος. Πέρας. Όχι ακόμα. Τώρα. Έληξε. 13-26 απορρίπτεται. 60 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Συμβασική 5 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 84 με 85 ψήφι υπέρ 84 και 85 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται, εγκρίνονται. 86-87 υπέρ εγκρίνονται. 89-90-91 ψήφι υπέρ κατά εγκρίνονται πάρα πολλοί συντάκτες λοιπόν. Πού να την απορρίψουμε. Συμβαστική αξιπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 98-103-104 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνονται. Προφορική τροπολογία 1 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 105 σε τμήματα. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 112 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 106, 107 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 108 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 109-110 υπέρ κατά αποχές έλεγχος. Πέρας. 15-27 απορρίπτονται. 111 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 113 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 114 υπέρ κατά αποχές δεκτή 115 υπέρ κατά αποχές δεκτή Συμβασκή 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 25 <clears throat> υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 26 υπέρ κατά αποχές δεκτή 27 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 28 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 29 υπέρ κατά αποχές έλεγχος 29, ναι. 30, υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 31 και 32, υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Δεκτές. 33, υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 34, υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Συμβαστική 3 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Στην 41 υπέρ κατά αποχές δεκτή, 42 υπέρ κατά αποχές δεκτή, 44 υπέρ κατά αποχές δεκτή, 46 υπέρ κατά αποχές απολύπτωται, 47 υπέρ κατά αποχές δεκτή, 49 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 50 και 51 υπέρ κατά αποχές δεκτή 52 υπέρ κατά αποχές δεκτή 1 υπέρ κατά αποχές δεκτή 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 4 υπέρ κατά αποχές δεκτή 6 υπέρ κατά αποχές δεκτή, 7 υπέρ κατά αποχές δεκτή, 8 και 9 που είναι ταυτόσιμες υπέρ κατά αποχές δεκτές, 10 και 11 υπέρ κατά αποχές δεκτές, 12-13 υπέρ κατά αποχές δεκτές, η ενα έχει εγκριθεί οπότε εκπίπτει 14, 15 υπέρ κατά αποχές δεκτή, 16 υπέρ κατά αποχές δεκτή, Προφορική τροποποίηση 5 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Συμβαστική 1 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Και τώρα η τελική ψηφοφορία. η ψηφοφορία. Πέρασε ψηφοφορίας. 37-4 και μία αποχή. Wir kommen zur Abstimmung des Berichts. Η εκθέση Κόβαλ, ο κύριο Κόβαλ δεν είναι παρόν, όμω ο κύριο Τάνεκ θα τον αντιμετωπίσει, θα τον αντικαταστήσει, συγγνώμη. Κατανοώ ότι έχουν γίνει κάποιε συμβαστικέ λύσει που έγιναν δεκτέ και μπορούμε να ψηφίσουμε κατευθείαν, κύριε Πρόεδρε. Πάμε. Συμβαστική 5 υπέρ. Κατά αποχέ δεκτή. Τροπολογία 78 υπέρ. Κατά αποχές <clears throat> δεκτή. 70... Α. <clears throat> υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω ότι απορρίπτεται, αλλά σε ελέγξουμε. παρακαλώ ιδιαίτερα το ΕΛΚ. Ο κύριο Σέβερν κάποιον έχει και τον υποστηρίζει μάλλον, λέει ο πρόεδρος. Λοιπόν, 80, όχι, έχουμε τη συμβαστική 6 του λέει η γραμματεία. Συμβαστική 6 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 84 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Συμβαστική 7 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Πάμε στην 93 υπέρ. 93. Έτσι γράφει εδώ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 98 λέει ο πρόεδρος. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 99. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 100 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 2.49 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 101 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 102 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 2.50, όχι. Συμβαστική 8 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 2.53 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 9 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 256 κάθετος 116 και 116 που είναι ταυτόσιμες. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτονται. 100... 117. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτονται. 118 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τσεκ. Έλεγχος στη δεύτερη τμήμα της 118. Πέρασε. εγκρίνεται. 2.57 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 2.58 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 119 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 10 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 133 υπέρ εγκρίνεται. Συμβαστική 11 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 12 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 1.51 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 152 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 2.62 υπέρ. Κατά αποχές 2,62 υπέρ. Κατά εγκρίνεται. 2,63 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 13 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 14 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 160 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 161 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστή 15 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστή 16 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 268. Φλέκενστάιν υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 17 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 20 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 198. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 199. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 200. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 201. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος. Abstimmung ist geschlossen. Απορρίπτεται. 202 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 269 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 206 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 210 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 211 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 272 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 214 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 215 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 273 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 216. Αποχές εγκρίνεται. 217 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Έλεγχος. 217 παρακαλώ. Έλεγχος. Ηλεκτρονικός. Πέρα εφορία. 15 υπέρ, 25 κατά, απορρίπτεται. 274 υπέρ. ...274 υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. 220 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 275 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 223 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 224 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 226 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 276 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Νομίζω ότι στην 200 26 έκανε ένα λάθος. Παρακαλώ να ψηφίσουμε ξανά την 226. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Νομίζω ότι είπα ότι απορρίπτεται. Λαθασμένα. 276 εγκρίθηκε. και 18 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Και τώρα περνάμε στην 231 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 232 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 19. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 278. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 233. Υπέρ. Την εγκρίναμε. Την 233. Υπέρ.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 32. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Νομίζω ότι εγκρίνεται, αλλά στο ελέγξουμε. Η 32, η 32. Ψηφίζουμε. Πέρα ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 34. Ναι, είναι λάθος. Καλύπτεται η 242. 34 λοιπόν, υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 35 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 3 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 44 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 45 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 46 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 47 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 48 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Η 48. 49-2-43 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 50 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 51 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 4 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 61. 62. 62. 62. 62 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 63 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Την 2.45 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Η 1 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Η 2 υπέρ. Σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές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 Να τα ψηφίσουμε όλα μαζί. μπλοκ. 11-17 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνονται. Και περνάμε στην τελική ηλεκτρονική ψηφοφορία. Έναρξη ψηφοφορίας. Antrag. Πέρασε. 36 ψήφοι υπέρ, 2 κατά, 2 αποχές. Κύριε Τάνοκ, ε, μεταβιβάστε στον εισηγητή τα συγχαρητήριά μας. Και τώρα περνάμε στο σχέδιο γνωμοδότησης για το πρωτόκολλο του Κιώτο. Υπέρ. Ελεκτρονικά, ελεκτρονικά. Για να καταγραφεί την ιστορία. τη ψηφοφορίας. 34 ψήφοι υπέρ, μία κατά, δύο αποχές. Και έτσι λοιπόν θα κάνουμε 15 λεπτά διάλειμμα. 10 λεπτά διάλειμμα. Και μετά θα έρθει ο Πιεδημόντ για να μας ε, παρουσιάσει τι υπόθηκε στο Συμβουλίο Υπουργών για το Εξωτερικών για την Ουκρανία. Πρόεδρε, να ενημερώσω τους συναδελφούς ότι από ό,τι φαίνεται οι Ρώσοι έχουν θέσει ε, τελεσίδικο για την ε, παράδοση της Κρυμαίας μέχρι αύριο στις 3. Αυτά αναφέρει το BBC και άλλα ειδησιογραφικά πρακτορία. Thank